Καλημέρα σας. 9 και 10 πάει η ώρα, οπότε είναι ώρα να ξεκινάμε. Τα πρακτικά των συντονιστών τα πήρατε μέσα στη νύχτα. Εάν μέχρι το τέλος συνεδρίασης δεν έχει κανείς καμία αντίρρηση ένσταση, θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών. Και ερχόμαστε στο πρώτο σημείο σήμερα το οποίο είχαμε αναβάλει από χτες, χειρεύει μια θέση αντιπροέδρου εδώ στην Επιτροπή μας και θα πρέπει να καλυφθεί. Διαπιστώνω και πάλι ότι στην αρχή της θητείας όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν για το πώς θα ε, κατανέμονται οι διάφορες θέσεις και τα οφήκια. Οι σοσιαλδημοκράτες ε, άφησαν μια θέση που είχαν στο Προεδρείο Γι' αυτό έχουμε πρόεδρο του ΕΛΚ, αντιπρόεδρο Πράσινο, ε, ελεύθερο, ε, γκούε και ε, της Ευρώπης για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Κανένα σοσιαλιστή και δημοκράτη. Αυτοί είναι οι κανόνες, αυτή είναι η συνένεση που επικράτησε εδώ στο Κοινοβούλιο και δεν βλέπω καμία αφορμή τώρα να σπάσει αυτή η συνένεση και να καταργηθεί. Ο νέος συνάδελφος από τη Φιλανδία ανήκει σε ένα κόμμα που δεν είναι ιδιαίτερα ευρωενθουσιώδης, αλλά αν είχε ε, βάλει υποψηφιότητα ένας σοσιαλδημοκράτης, ε, Φιλανδός, θα ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες. Γιατί και αυτοί αρνήθηκαν τις ενισχύσεις για την Ελλάδα και τη Βορτογαλία. Λοιπόν, είτε έχουμε κανόνες και ε, θα καλωσορίσουμε το συνάδελφο ε, διαβοής, είτε έξι συνάδελφοι θα εγερθούν και θα ζητήσουν μυστική ψηφοφορία για την κάλυψη αυτής της θέσης. Θέλετε μυστική ψηφοφορία? Εσύ, χάνω, όχι βέβαια, η Μαρία Μπαντία. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν χρειάζεται με μυστική ψηφοφορία διανατάσσεως του χειρός και τελειώνει η υπόθεση για μυστική. Έκανε κάποια σχόλια η πρόεδρος σε σχέση με κάποια κόμματα και εγώ θα ήθελα πολύ σύντομα να αναφερθώ σε αυτά, μου επιτρέπετε. Είναι γεγονός ότι σε κάποια θέματα ορισμένα κόμματα είχαν αντίστοιχη στάση στην προεκλογική εκστρατεία. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονούμε ότι και σε άλλα θέματα όμω ρατσισμού και ξενοφοβία, απέχουμε πόρο από το κόμμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν θα μπούμε τώρα σε τέτοια συζήτηση. Ήθελα να το ξεκαθαρίσω και να ζητήσω από την Πρόεδρο Συμφωνία να ψηφίσουμε διανατάσεις της χειρό. Δυστυχώ δεν γίνεται αυτό, δεν προβλέπεται είτε διαβοή είτε με μυστική ψηφοφορία. Διανατάσεω δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Και εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω. Μαρία. Μαρία Μπαντία. Δεν έχω εδώ τα χαρτιά μου, δεν ξέρω αν αυτό που μας λέτε ισχύει, αλλά σας εμπιστεύομαι, είμαι υποχρεωμένη άλλωστε. Κάθε φορά που ζητήθηκε εδώ ψηφοφορία γινότανε. Άλλο είναι μυστική ψηφοφορία. Όταν ζητάμε με ηλεκτρονική κάρτα, για πρώτη φορά μου λένε ότι δεν μπορώ να ζητήσω ψηφοφορία δυνατά σε οσχυρό και πρέπει να γίνει διαβοή. Τότε γιατί ψηφίζουμε. Γιατί μας ε, το υποβάλλετε στην κρίση μας αν είναι διαβοής. Δεν το ξέρω. Σας εμπιστεύομαι, σας πιστεύω αυτό που λέτε, αλλά θα ήθελα παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά ότι θέλω να το επαληθεύσω, γιατί μου φαίνεται η κατάσταση λίγο μυστήρια. Ε, Μαρία. Αυτό το λέει ρητά στο άρθρο 191 εδάφιο 2 σε σχέση με ε, τον αριθμό των υποψηφίων για μία θέση που χειρεύει. Μπορεί να γίνει διαβοής. Όταν δεν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφοι ή εάν το ζητήσει το 1 έκτο, το 1 έκτο των μελών, της Επιτροπής η ψηφοφορία αυτή διεξάγεται μυστικά. Δηλαδή, αν βρεις έξι μέλη να γερθούν, να το ζητήσουν, εν πάση περιπτώσει, θα ψηφίσουμε με μυστική ψηφοφορία. Μαρία Μπαντίας. Δεν μ' αρέσει που χάνουμε χρόνο με αυτό το πράγμα εξαιτία μου, αλλά για να το διευκρινίσουμε. Λέτε ότι σε περίπτωση που υπάρχει άλλο υποψήφιο μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορούμε και εμεί να κατεβάσουμε υποψήφιο και έχουμε δύο αμέσω αμέσω. Εγώ δεν ξέρω από τέτοια πράγματα, δεν σκαμπάζω από νόμους και κανονισμούς, αλλά θα ήθελα και ήλπιζα δημοκρατικά, αν υπάρχει μια διαφωνία κάπου, σε αυτό το κόμμα. Ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για πρόσωπα, κυρία Πρόεδρε, όλοι παρόντες εδώ. Να μπορεί ο καθένας να δείξει πώς ψηφίζει, να συμφωνεί ή όχι, και τίποτα παραπάνω. Δεν μπορώ παρά να σας ξαναδιαβάσω αυτά που ορίζει ο κανονισμός. Κατόπιν ετήσεως εκτίματος μάλλον ενό έκτου των μελών γίνεται μυστική ψηφοφορία. Αν βρείτε τώρα έξι μέλη που ζητούν μυστική ψηφοφορία μπορούμε να το πράξουμε. Ζητάς αυτό να γίνει μυστική ψηφοφορία. Θέλεις μυστική ψηφοφορία στα αγγλικά και στα γερμανικά η πρόεδρος. Yes. So, who is in favor... Μάλιστα. Ποιος είναι υπέρ της μυστικής ψηφοφορίας. Έξι χρειάζονται. Τέσσερις. Κατά. Δεν φτάνουν οι τέσσερις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω τους κατά καθόλου. Έξι χρειάζεται. Προχωράμε. <laughs> Λοιπόν, Παρακαλώ τους συναδέλφους ε, να ε, αντικαταστήσουμε το, το συνάδελφο Σόν με τον άλλο συνάδελφο που δεν θυμάμαι το όνομά του, εν περιπτώσει, διαβοής. Ελάτε, να καθίσετε δίπλα στον κύριο Μπίσκι που είναι η θέση σας. Λοιπόν, πάει το πρώτο θέμα. Ερχόμαστε στο σημείο 10 της μέσης διάταξης η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2012. Όχι στη θέση του κύριου Μπίσκι, δίπλα στον κύριο Μπίσκι. Τι είπατε εσείς. Είπατε στη θέση του κυρίου Μπίσκι. Όχι κυρία μου, είπα δίπλα στη θέση του κυρίου Μπίσκι. Θεέ μου, τι το κάναμε εδώ πέρα. <laughs> Πάντως όχι Επιτροπή Πολιτισμού. Έχω την εντύπωση. Σημείο 10. Ο εισηγητή είναι ο κύριος Λόκεγκαρτ για τον προπολογισμό του 2012. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι η δεύτερη χρονιά που διατελώ εισηγητή για τον προπολογισμό τη επιτροπή μας. Πέρσι καταφέραμε να αφήσουμε το στίγμα μας ε, στον προπολογισμό στην τελική εκδοχή για τη διαβίου ε, μάθηση. Ε, δεν ήταν καμιά φανταστική επίδοση, αλλά καλό είναι και αυτό. Ορισμένοι λέγουν ότι δεν αρκεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, αλλά και οι δύο απόψεις έχουν δίκιο. Η λιτότητα ε, κυριάρχησε πέρσι και ήταν η κεντρική ιδέα στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, όπως και φέτος άλλωστε. Και φέτος θα πρέπει να περιοριστούμε και να σεβαστούμε ε, τους δύσκολους ε, καιρούς που περνούν από δημοσιονομικής απόψεως στα κράτη με σκληρές οι δημοσιονομικές συνθήκες. Από την άλλη θα πρέπει να αγωνιστούμε για αύξηση των ε, κονδυλίων του προπολογισμού. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι το έχει ε, ορίσει αυτό το δίλημα. Ωραία. Είναι μια λεπτή ιστοροπία όπου χρειάζεται να συνδυαστεί η λιτότητα με μέτρα που θα ε, ενισχύσουν και θα τονώσουν την ανάπτυξη. Θα θυμάστε ότι έχω πει και στο παρελθόν ότι φέτος θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεντρωμένοι με στόχους, να ξέρουμε τι προτεραιότητες έχουμε και να επιμείνουμε να μας δώσουν τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό χρειάζονται μεταφορές πιστώσεων σε κάποιες σημαντικές πιστώσεις ουσιαστικές για μας για τη στρατηγική του 2020. Για ποιο λόγο τα λέω όλα αυτά. Διότι για να πετύχει η στρατηγική αυτή χρειάζεται ε, τους απαραίτητους πόρους και θα πρέπει να γίνουν οι σωστές επενδύσεις. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν έξτρα πόρους για να επενδύσουν στην παιδεία, για παράδειγμα, και είναι φαύλος κύκλος αυτό τελικά. Εάν δεν επενδύουμε σήμερα στην παιδεία, τότε δεν πρόκειται να ε, έχουμε θέσει απασχόλησης και ανάπτυξη στο μέλλον. Ευτυχώς ο Γενικός συγητή για τον Προπολογισμό, η Συγήτρια μάλλον το 2012, η κυρία Μπαλζάνη, η σοσιαλίστρια, ε, ε, είναι προσιλωμένη στους στόχους της στρατηγικής 2020 και πιστεύω ότι ε, θα υποστηρίξει την αύξηση της πρικοδότησης της διαβίου μάθησης και νομίζω ότι θα είναι από τις προτεραιότητές μας αυτό για φέτος. Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Συμβούλιο δεν κατάφερε να αυξήσει τα κονδύλια για την Ευρώπη του 2020. 4,5% προτείνεται για τη διαβιομάθηση, αλλά αυτό ε, ρέει από το πολιετές πλαίσιο του προγράμματος και τον πληθωρισμό. Δηλαδή ονομαστική αύξηση, αλλά ουσιαστική όχι. Μία μόνο γραμμή του προϋπολογισμού στο σχέδιο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρικοδοτείται επιπλέον, που είναι νεολαία σε δράση, 5 εκατομμύρια επιπλέον, καλό είναι αυτό βεβαίως αφού συνεισφέρει και στη γενικότερη στρατηγική για το 2020. Δυστυχώς όπως σας είπα είναι η μοναδική αύξηση κονδυλίου φέτος για τα θέματα που μας αφορούν. Θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα χρήματα για την παιδεία που είναι πραγματικά το κλειδί παντού ε, στη στρατηγική μας. Αυτά ε, γενικά. Να σας πω δύο λόγια για τη διαδικασία. Πέρυσι ήταν η πρώτη φορά με την ε, πρώτη ετήσια δημοσιονομική διαδικασία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, βασικά ένα μπάχαλο ήταν. Κατέψαμε να χάσουμε και τα Χριστούγεννα μας στις διακοπές. Τελευταία ώρα συμφωνήσαμε στο παραπέντε. Φέτος, μία από τα ίδια. Η θέση του Συμβουλίου θα έρθει πολύ αργά, τον Ιούλιο κάπου, στα τέλη Ιουλίου και περισσότεροι από εμά θα έχουμε φύγει ε, για διακοπές και συντονιστές της Επιτροπής μας ε, αποφασίσαμε να ψηφίσουμε στις 14 Ιουλίου ε, τις τροπολογίες μας και να τις καταθέσουμε και να τις ψηφίσουμε στα αγγλικά γιατί δεν θα υπάρχει και χρόνος για μετάφραση. Ως εισηγητής της Επιτροπής μας θα ζητήσω ε, γενική εντολή οριζόντια για να διαπραγματευτώ το Σεπτέμβριο και για το σχέδιο προϋπολογισμού αν θα έχει προτείνει περικοπές στο Συμβούλιο. Στην πράξη τι σημαίνει αυτό, ότι τον Ιούνιο θα κάνουμε μια γενική συζήτηση στη συνεδρίαση μας για το σχέδιο προϋπολογισμού, θα σας καταθέσω τις πρωτο... τροπολογίες μου και μετά θα οριστεί η προθεσμία κατάσταση τροπολογιών για όλες τις τροπολογίες του προϋπολογισμού. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο μπορεί να κάνει περικοπές στο σχέδιο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν θέλετε τα ποσά που έχει προτείνει η Επιτροπή και τα περικόψει στο Συμβούλιο, δεν χρειάζονται νέες τροπολογίες. Ε, θα με εξουδοτήσετε, θα έχω την εντολή να το κάνω εγώ εξ ονόματό σα το Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα κάνετε τροπολογίες στα αγγλικά, όπω σας είπα. Θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μα τον Ιούλιο και ε, μετά το Σεπτέμβριο όταν θα έχουμε τα αριθμητικά στοιχεία του ε, Συμβουλίου. Δεν ξέρω, το είχατε καταλάβει. Σας φαίνεται σαφές, τουλάχιστον προσπάθησα να σας το εξηγήσω όπως μπορούσα, όσο καλύτερα μπορούσα. Σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό θα είναι σύντομο κείμενο όπως και πέρσι, 5-6 παράγραφοι. Θα σας φέρω στις 14 Ιουλίου ένα προσχέδιο και στις 5 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Τέλος, Δύο λόγια για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Η Επιτροπή Προϋπολογισμού ε, ζήτησε ε, αναδιατάξει τα κονδύλια, όπως ξέρετε. Η εσωτερική προθεσμία εδώ στην Επιτροπή μας ήταν η τρίτη που μας πέρασε. Η Επιτροπή λοιπόν, της Γραμματείας θα τα στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα επανέλθουν Προσέξτε ότι θα πρέπει να ε, υποβληθούν ε, σωστά αυτές οι δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα ως τροπολογίες στον προπολογισμό ακόμα και αν έχετε στείλει τα σχετικά έγγραφα στην Επιτροπή μας, στη Γραμματεία. Τέλος, η δική μου θέση, όπως έχω ξαναπεί, είναι ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να αυξηθεί η υπηκοδότηση στη διαβίου μάθηση. Αν θέλουμε να φτάσουμε κάπου πρέπει να έχουμε σαφείς στόχους και να εστιαζόμαστε να εστιάζουμε συγγνώμη σε αυτούς. Επίσης για τον αθλητισμό υπάρχουν μερικά ε, καλά πιλωτικά προγράμματα και όταν θα έχουμε τις προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθίσουμε να το συζητήσουμε για να συμφωνήσουμε σε μία ή δύο το πολύ ε, που θα έχουν την υποστήριξη ολόκληρης της Επιτροπής Πολιτισμού. Αυτά εισαγωγικά. Όσο μεγαλύτερη η υποστήριξη, τόσο μεγαλύτερε είναι και οι πιθανότητες ε, να ε, επικρατήσουμε στο τέλος και να στείλουμε σαφέ μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για φιλόδοξο πρόγραμμα και για τον αθλητισμό. Όλοι φανταζόμαστε είμαστε υπέρ. Δεν θα αναφερθώ σε περαιτέρω προγράμματα τώρα, απλώ να μην δεχτούμε καμία περικοπή στα κονδύλια που μας αφορούν. Αν δείτε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι στιγμής, νομίζω ότι εγγράφεται και στη δική μας γραμμή, οι δικές μας πιστώσεις σαφέστατα προσθέτουν ευρωπαϊκή αξία και συνεισφέρουν ε, στη στρατηγική 2020 και στο κάτω-κάτω είναι και δημοφιλή προγράμματα και δράσεις ε, στον πληθυσμό. Νομίζω λοιπόν έχουμε κάθε πιθανότητα να επιτύχουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για άλλη μια φορά θα ήθελα να επανέλθω και να πω ότι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι και συμφωνώ το ότι θα πρέπει να προχωρήσει και να υποστηριχθεί. Δεν ξέρουμε ποιες αλλαγές θα επιφέρονται από το Συμβούλιο. Θα ασχοληθούμε όμως με αυτές όταν θα γίνουν. Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι ή το Συμβούλιο, ε, κατά πόσον τώρα αυτό θα είναι θέμα αξιοπιστίας, πρέπει να δοθούν περισσότερα κονδύλια για τους επιμέρους τομείς, ιδιαίτερα για την διαβίου μάθηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω, έχω μια παρατήρηση να κάνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές ερωτήσεις για ειδικέ εκδηλώσεις, special events. Οι ειδικέ αυτές έκτακτες εκδηλώσεις πολλές φορές ε, βρίσκονται στον τομέα του αθλητισμού. Δεν πιστεύω όμως ότι την προσέγγιση για τον αθλητισμό που είναι τόσο περιορισμένη και ουσιαστικά και δεν υφίσταται γιατί προσπαθούμε να συλλέξουμε κονδύλια έστω. Αυτή η προσέγγιση για τον αθλητισμό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ειδικέ έκτακτες εκδηλώσεις. Αυτή η προσέγγιση για τον αθλητισμό πρέπει να εντάσσει αυτά τα οποία ω πιλωτικά προγράμματα έχουν συλληφθεί, έχουν επινοηθεί και μετά να ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα για τον αθλητισμό. Οι έκτακτες εκδηλώσεις και πολλές φορές αφορούν βέβαια τον αθλητισμό πρέπει υπό το ειδικό κονδύλιο που υφίσταται για έκτακτες εκδηλώσεις να ενταχθούν, σε αυτό να ενταχθούν. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω αυτό στους συναδέλφους. <clears throat> Αναφέρθηκαν οι αθλητικές ε, δραστηριότητες ε, που όπως η ε, ειδική Ολυμπιακή κύριε Τάκολα ή τα, οι χειμερινοί αγώνες νέων στο Ινσπρουκ. Όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από τα πιλωτικά προγράμματα. Το πιλωτικό πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο έχει πιο μακροπρόθεσμη, ας το πω έτσι, πιο μακροπρόθεσμο χρονοορίζοντα και δεν είναι εφήμερη εκδήλωση. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να το δούμε. Φυσικά μπορούμε να διαβιβάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο αυτά τα οποία είναι αυθεντικό πιλωτικό πρόγραμμα έχουν συλλεγεί κάποια στοιχεία, έτσι δεν είναι. Χθε ή προχθέ είχαμε την καταληκτική προθεσμία. Η Γραμματεία θα υποβάλει αυτές τις ε, προτάσεις. Θα δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιο είναι το πιο κατάλληλο για να μπορέσει να, να υλοποιηθεί. Και αυτό σε σχέση με τις προτάσεις ε, που θα έχουν φιλτραριστεί πιο πριν. Δεν είναι δυνατόν παντός του επιστητού να υποβάλλονται προτάσεις. Είναι λοιπόν θετικό έτσι να εξετάσουμε αυτό το θέμα για τις ειδικέ εκδηλώσεις αυτή, αυτό το θέμα είναι ξεχωριστή ιστορία. Πρέπει ξεχωριστά να συζητήσουμε για αυτό το θέμα για το σχέδιο προϋπολογισμού όταν θα έρθει η ώρα. Θα υπάρξουν αθλητικές εκδηλώσεις που ίσως θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Ο κύριος Μπέρετ συνάδελφος ζήτησε τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε κύριο Μπελέτ. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, υποστηρίζω αυτά που πρότεινε ο εισηγητής. Η πολιτική μου ομάδα σε μεγάλο βαθμό τον υποστηρίζει. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικά μας βρίσκει σύμφωνο, γιατί ε, υπάρχουν κάποια θέματα ζωτικής σημασίας για μα και αυτά τα αναφέρατε. Είναι στρατηγική το 2020. Θα πρέπει να παραμείνει η χρηματοδότηση για το, ε, τα μίντια, για τι ανταλλαγέ νέων, για τη διαβίου μάθηση. Γενικά ε, συμφωνούμε και θα πρέπει να επενδύουμε πολύ περισσότερο σε αυτούς τους τομείς για να φτάσουμε και στους στόχους ε, του 2020. Ε, νέα προσόντα, νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας, αυτό ε, προβλέπεται και καλό είναι να διατηρηθεί η χρηματοδότηση. Λυπάμαι πάρα πολύ που τώρα δεν έχουμε χρήματα για τον προπολογισμό εκτός από τις προπαρασκευιστικές δράσει. Ελπίζω να βρούμε τα κονδύλια από αλλού. Συμφωνώ απολύτως με την Πρόεδρο. Για να στείλουμε ένα μήνυμα, μπορεί να είναι νωρί βέβαια ακόμα, για την πολυετή μα προετοιμασία. Προετοιμαζόμαστε αυτόν τον καιρό. Κυκλοφορούν διάφορε φήμε στου διαδρόμου και νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε ήδη από τώρα ένα πλήρες ε, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τον αθλητισμό και είναι και αποτελεσματικό εργαλείο και μέσο για τη διασυνορική συνεργασία και για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνοχή. Και ξέρετε φυσικά ότι ο αθλητισμός καταπολεμά και διάφορα προβλήματα υγείας τα προλαμβάνει μάλλον. Επίσης, υπάρχουν διάφορες δομές που λειτουργούν ήδη. Ε, διάφορα προγράμματα δικά μας στο νεολαία σε δράση, ε, διαβίου μάθηση και θα πρέπει ε, να τα προωθήσουμε και να τα συνεχίσουμε. Δηλαδή κάποιες δομές που λειτουργούν σωστά θα πρέπει να συνεχίζονται και με τη σωστή χρηματοδότηση. Γενικά πάντως θα ήθελα να πω ότι η ομάδα μας υποστηρίζει την πρόταση που έχουμε επιτάπητος από πλευρά του μας μικρόφωνο. Κυρία Παλιαδέλη, παρακαλώ. Φράου ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, καταρχήν να ομολογήσω, να δηλώσω ότι νιώθω ιδιαίτερα ασφαλής ότι γενικό, ε, ο ραπορτέρ για την εισηγήτρια για τον συνολικό προϋπολογισμό είναι η κυρία Μπαλτσάνη και επίσης ασφαλής ότι για δεύτερη χρονιά φέτος η ε, εισηγητής μας από, στην Επιτροπή Πολιτισμού ε, είναι ο κύριος ε, Λόκεγκαρτ. Ε, για μένα είναι η πρώτη φορά που μετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Ομολογώ ότι δεν είναι όλα πολύ το σαφή, αλλά έχοντας μια γνώση από δημοσιονομική πολιτική στην χώρα μου, σας δηλώνω ότι θα κάνω κάθε προσπάθεια προκειμένου να υπηρετηθούν οι στόχοι τους οποίους ανέφεραν και οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι και τους οποίους συμφωνώ, οποίους συμφωνώ απόλυτα. Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα όταν διαπίστωσα ότι ο τομέα 3, στον οποίο υπάγεται ο πολιτισμό και η εκπαίδευση, έχει συνολικά το 1,2% του συνολικού προπολογισμού και η ηθαγένεια, στην οποία ακόμη ειδικότερα υπαγόμαστε, έχει μόλι το 0,5% του, του συνολικού προπολογισμού. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Βεβαίω όχι τώρα, στην περίοδο που έχουμε αυτή την τεράστια ε, οικονομική κρίση και ως Ελληνίδα το καταλαβαίνετε ίσως περισσότερο από όλους ότι είμαι ευαισθητοποιημένη στο σημείο αυτό αλλά να μην ξεχνούμε ότι <clears throat> τα θέματα τα οποία μας απασχολούν στην Επιτροπή στην ουσία ε, μπορούν να γίνουν ανταποδοτικά δηλαδή και ο πολιτισμός και η εκπαίδευση και ο αθλητισμός ε, είναι ανταποδοτικά από μόνα τους επομένως πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε προσπάθειες προκειμένου να αυξήσουμε ε, κονδύλια ε, σε ορισμένους τουλάχιστον ε, τομείς. Είναι σημαντικό ότι ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα της Ευρώπης και τα πιο πετυχημένα, το Εράσμους, τώρα το Εράσμους Μούντους και το πρόγραμμα για τη διαβίου μάθηση δεν υφίστανται μειώσεις αλλά έστω και μικρές αυξήσεις και χαίρομαι ότι η νεολαία σε δράση έχει ε, πάρει περισσότερα χρήματα από την περασμένη ε, χρονιά λόγω του γεγονότος ότι εντάσσεται στην, ευρωπαϊκή, στην εμβληματική πρωτοβουλία νεολαία σε Ε, λυπούμε ότι το media, ε, το πρόγραμμα Media θα μπορούσαν, δεν έχουν δεχτεί τόσες πολλές, δεν, δεν έχει δεχτεί αύξηση και ειλικρινά επειδή εντάσσεται σε αυτό και η τηλεόραση και ο, πολιτι... και ο κινηματογράφος ο ευρωπαϊκός. Εδώ θα πρέπει να βρούμε τρόπους κάποια στιγμή να τους ενισχύσουμε γιατί κακά τα ψέματα έχουμε δει ότι γενικά ο πολιτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και βεβαίως μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Ε, επομένως, ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Πιστεύω βαθύτατα ότι ο πολιτισμός είναι ένα τομέα και η εκπαίδευση για το μέλλον της Ευρώπης και ο πολιτισμός άμεσα Επομένως, ό,τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, έστω με αυτά τα χρήματα, προκειμένου να, να, να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους προγράμματα και να αξιοποιήσουν τα χρήματα, τα λιγοστά χρήματα που διατίθενται, θα είναι για το καλό της, Ευρώπης, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τη. Ε, ελπίζω ότι θα συνεργαστώ πολύ καλά με τον κύριο Λόκιγκαρτ ε, προκειμένου να πετύχουμε τους κεντρικούς στόχους όπως περιέγραψε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, Ευχαριστώ. Φύσας παρακαλώ. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο συνάδελφο Νόκεγκαντ για το έργο που επιτελεί σε αυτό το θέμα που είναι τόσο θα έλεγα ε, θέμα δύσκολο και ευχαριστούμε για αυτή την προσπάθεια για τη διασφάλιση κονδυλίων. Δεν είχα την ευκαιρία να τα δω όλα σε βάθος παρότι το ήθελα θα μπορεί να υπάρχουν προτάσεις που πρέπει να προαχθούν. Θέλω να τονίσω αυτό το οποίο είπε η Πρόεδρος σε σχέση με τις προτάσεις για τον αθλητισμό. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνουν δεκτά προγράμματα πιλότη, πιλότ που θα έχουν αιτήσιο χαρακτήρα. Γι' αυτό υπάρχει ήδη ένα κονδύλιο ξεχωριστό στον προϋπολογισμό για έκτακτες αιτήσιες εκδηλώσεις αυτό το γεγονός, αυτή η εκδήλωση στη Λιθουανία για παράδειγμα. Και θα έπρεπε να πούμε ότι θα πρέπει σε αυτό το κονδύλιο να στραφούν και να αντληθούν από εκεί κονδύλια και όχι από ένα πρόγραμμα πιλότου, πιλωτικό. Τα προγράμματα τα πιλωτικά πρέπει και όταν θα έχουμε περισσότερα χρήματα 2014 θα πρέπει εφόσον θα μπορεί να είναι ενδιαφέροντα, τότε να μπορούν να ενταθούν στον γενικό προϋπολογισμό τέτοιου είδους ε, εκδηλώσεις, αλλά όχι σε σχέση με τα πιλωτικά προγράμματα. Στο ειδικό κονδύλιο για τις ετήσιες εκδηλώσεις λοιπόν. Και έτσι ευχαριστώ τον κύριο Λόκ για την προσπάθεια που κάνει να έχουμε τον, την καλύτερη δυνατή λύση από πλευρά κονδυλίων. Ευχαριστώ. Χάνω Τάκουλα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ από πλευράς μου μπορώ να πω και να διαπιστώσω ότι με ικανοποιεί και είμαι και υπερήφανος για το ότι ο κύριος Λόκεγκορντ εργάστηκε τόσο καλά. Δεν έχω παρατηρήσεις. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η γραμμή που μας παρουσίασε, μας πρότεινε η πρόεδρός μας όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα, είναι κάτι επί της οποίας αυτής πρότασης συμφωνώ. Αυτά είναι τα κέντρα βάρους που θα έπρεπε να έχουμε όταν ακριβώς ε, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία ισχνότητας κονδυλίων. Όσον αφορά τις έκτακτες εκδηλώσεις, ειδικές εκδηλώσεις, θα έπρεπε με κάποιο ειδικό τρόπο να διασφαλίσουμε ώστε να πετύχουμε από πλευρά προπολογισμού ώστε αυτές οι δύο εκδηλώσεις ε, που ετήσια ε, σε τακτά διαστήματα θα πρέπει να υποστηρίζονται οι ειδικοί Ολυμπιακοί αγώνε για άτομα με ειδικέ ανάγκες ή, ε, ή τα οι αθλητικές εκδηλώσεις για τους νέους στη Ρουμανία. Αυτές οι ε, που παραδοσιακά υποστηρίζαμε να μπορέσουν ε, να τύχουν υποστήριξη κατά κάποιο τρόπο. Κρίμα είναι ότι δεν έχει ξεχωριστό προϋπολογισμό ο αθλητισμός. Η ιδανική περίπτωση αυτή θα ήταν να υπήρχε ένας ειδικό προπολογισμό για τις εκδηλώσεις ε, στο πλαίσιο του αθλητισμού. Εφόσον δεν γίνεται αυτό και δεν διασφαλίζεται θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Είναι εκδηλώσεις που έχουν ε, σημασία και σπουδαιότητα όταν πρόκειται για το δικό μας ρόλο, για την καταπολέμηση του ρατσισμού και την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και υπέρ των, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να αποδείξουμε και να σηματοδοτήσουμε ότι κάθε νέος, κάθε παιδί έχει δικαίωμα στον αθλητισμό και να μπορεί να ασχολείται και να χαίρεται ε, ασχολούμενο με τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός είναι κάτι που μπορεί να προαγάγει την συνεργασία και πρέπει να υποστηριχθεί. Αυτή είναι η τομή που θα έπρεπε να τονίσουμε και πρέπει στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή να βρούμε κάποιο τρόπο να υποστηρίξουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Καταρχήν συμφωνώ με την Πρόεδρο σε αυτά που είπε. Πρέπει να έχουμε στα πιλωτικά Ευχαριστώ. στην δική μας αυτή ε, πραγματικότητα όταν έρχεται η ώρα να δούμε τα κονδύλια και να δούμε τι μπορεί να γίνει δεν είναι η σημαντική αύξηση εκείνη που ζητάμε. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να υπάρχουν τέτοιου είδους αυξήσεις άσχετα από την οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε πρέπει πολύ δύσκολες ε, σκληρές αποφάσεις να λαμβάνονται σε αυτή τη συγκυρία για περικοπές ε, και αυτή είναι η κατάσταση. Απευθύνω έκκληση να δουν τα μέλη την απόφαση του Συμβουλίου να επανεξεταστεί η ανάγκη που υπάρχει σε σχέση με τα κράτη-μέλη να υπάρξουν προσαρμογές ε, σε σχέση με αυτά τα οποία κάνουν και οι εθνικές κυβέρνησεις δημοσιονομικά. Όμως κατ' εκτίμηση ως θέμα αρχής πρέπει σε σχέση με τα θέματα πολιτισμού εμείς ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσουμε την αξία που θα επιτυγχάνουμε από τα χρήματα, τα κονδύλια που θα διαθέτουμε. Πρέπει να υπάρξει ιεράρχηση για αυτούς τους τομείς που θέλουμε να δράσουμε και να διασφαλίσουμε ότι οι πρωτοβουλίε που θα χρηματοδοτούμε θα είναι σωστέ και θα υπάρχει πρόσθετη αξία. Αυτό θέλω να ενθαρρύνω του συναδέλφου να κοιτάξουν και σε σχέση με αύξηση κονδυλίων. Υπάρχουν αυξημένε προσδοκίε φυσικά στον τομέα του αθλητισμού και ίσως θα πρέπει να δούμε αν αυτό μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα. Πρέπει να υπάρξει ιεράρχηση λοιπόν των σωστών προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Έχω την εξή ερώτηση προς τον κύριο Μπερνάρ Νάουστα. Α, εσείς παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βλέπω ευρία υποστήριξη για την πρόταση της Κομισιόν που είναι όντως ε, ε, ένα ρεαλιστικό μείγμα λιτότητας και προσπάθειας εκεί που μπορούμε να στηρίξουμε ε, τα προγράμματα αυτής της Επιτροπής. Είδαμε ότι παραμείναμε στον πολιετή σχεδιασμό για τα περισσότερα προγράμματα δεν υπάρχουν περικοπές στο πολιετές πρόγραμμα, ενώ αν δείτε άλλους τομείς συμβαίνει αυτό φέτος. Εδώ όχι. Και σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, Youth in Action, όπως αναφέρθηκε, προσθέσαμε και 5 εκατομμύρια, γιατί διαφορετικά θα είχαμε πολύ περίεργο προφίλ λόγω των αυξήσεων στα προηγούμενα χρόνια. Θα βλέπαμε εδώ μέσα στο πλαίσιο του πολιετούς προγράμματος μείωση, που θα, πράγμα που θα έδινε λάθος μήνυμα. Γι' αυτό και το αυξήσαμε κατά 5 εκατομμύρια ώστε να έχουμε μια διαρκή αύξηση. Όπως σας είπα, ο γενικός προπολογισμό είναι ρεαλιστικός και γι' αυτό και καλωσορίζω αυτά που άκουσα εδώ. Ότι σε περίπτωση που το Συμβούλιο προσπαθήσει να περικόψει κάποιες από αυτές τις γραμμές θα πρέπει να μας στηρίξετε και να επαναφέρετε τα ποσά τα οποία εμείς θεωρούμε ως μίνιμουμ ποσά. Επίσης αναφέρατε ο κύριος Λόκεγκάρντ κυρίως ότι στοχεύει στην ε, διαβίου κατά ε, ε, μάθηση εκεί να υπάρξει κάποια αύξηση. Νομίζω ότι είναι καλός ο στόχος όπως και το Youth in Action. γιατί έχει άμεσες επιπτώσεις σε διάφορους από τους ε, τομείς ε, που θεωρούμε σημαντικούς και γι' αυτό και θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο. Στρεφόμενοι στο θέμα του αθλητισμού, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για την Επιτροπή τούτη ως συνήθως και να καλωσορίσω επίσης τα όσα είπατε κυρία Πρόεδρε ότι δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε τους λιγοστούς πόρους σε πραγματικού και σε δράσεις που έχουν που φαίνεται ότι κάτι θα αλλάξουν πιο μακροπρόθεσμα στον τομέα γιατί με μονομένες δράσεις Εντάξει, πάντοτε μπορεί κανείς να τις υποστηρίξει, αλλά τελικά δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα της ίδιας, ε, τον ίδιο αντίκτυπο όπως οι πιλωτικές δράσεις. Γι' αυτό και θα θέλαμε να έχουμε μια συνεργασία μαζί σας, να βασιστούμε στις δράσεις που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, να δούμε τι είδους δράσεις θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε για να μέχρι το 2014 που σίγουρα θα έχουμε πιο μόνιμα προγράμματα για τον αθλητισμό καθώς οι αποφάσεις ακόμα δεν έχουν ληφθεί για όλα αυτά, όπως ξέρετε. Θα το δείτε σε κανένα μήνα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Καλωσορίζω και την υποστήριξη για τα περισσότερα προγράμματα, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να εστιάζουμε σε διάφορα πράγματα. Η βασική γραμμή λοιπόν για τον αθλητισμό και την διαβίου μάθηση είναι σε σωστός προσανατολισμός. Ευχαριστώ. Λόκεγκάρντ. Κάποια σχόλια για τα όσα ήδη υπόθηκαν. Φυσικά και στηρίζω επίσης τη στρατηγική να εστιάσουμε στην μακροπρόθεσμη ε, αξία των ε, προγραμμάτων και θα ήθελα να προσθέσω στα όσα είπαν οι συνάδελφοι ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποια από αυτά τα γεγονότα, να βρούμε και κάποια στέγη για όλα αυτά. Τα δύο τελευταία χρόνια πριν να μπούμε στο επόμενο πολιετές πρόγραμμα, ο χρόνος τελειώνει για τα τις, τις, τις υπάρχουσες δράσεις για τον αθλητισμό μας τον τελευταίο χρόνο και είναι προφανές κατά τη γνώμη μου ότι χρειάζεται κάτι παρόμοιο ε, που θα πρέπει να λειτουργήσει για τα τελευταία δύο χρόνια πριν να ξεκινήσουμε με το ε, οικονομικό μας ε, τον νέο μάλλον οικονομικό προσανατολισμό. Φαντάζομαι ότι κάτι θα μπορέσουμε να βρούμε, θα τα καταφέρουμε. Ε, ευτυχώς υπάρχει ευρεία συνένεση για τη γραμμή που ακολουθούμε και αυτό μας ικανοποιεί. Σας υπόσχομαι ότι θα δουλέψω πολύ σκληρά για να <laughs> βρούμε τα χρήματα. Τέλος, μια υπηρεσιακή πληροφορία. Δεν ανέφερα τα περιθώρια φέτος. Το 1α είναι 150 εκατομμύρια και στη 3β το ίδιο όπως και πέρυσι, δηλαδή 15 εκατομμύρια, που δεν είναι πολλά. Αλλά θα δούμε τι θα καταφέρουμε με αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Λόκεγκαρτ, να επανέλθω έχοντας αυτό το εγγραφό δημοσιονομική διαδικασία 2012 της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ε, για τον Πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το έγγραφο. Μπορεί κανείς να δει ποια είναι τα διαφορετικά κονδύλια πρώτο. Δεύτερο, μπορεί κανείς να δει ποια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και περιγράφονται όλα αυτά. Και έτσι μπορεί κανείς να δουλέψει με βάση αυτό το έγγραφο. Μπορεί επίσης να δει κανείς τι γίνεται από πλευράς Επιτροπής Προϋπολογισμών, τι έχουν εντάξει στο έγγραφό τους ε, για την διαβίου μάθηση. Είναι λοιπόν χρήσιμο να το έχει κανείς και να το κρατήσει αυτό μέχρι και τον επόμενο προϋπολογισμό, να δούμε ποιε είναι οι προοπτικές για αυτά τα θέματα. Ήθελα μόνο να σας ευαισθητοποιήσω γι' αυτό και έτσι χρειάστηκε και εγώ να αντιληφθώ ότι έπρεπε να σας το πω γιατί είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Από την άλλη πλευρά, σε σχέση με την κυρία Μακλάκιν, θα ήθελα να πω δύο λόγια στα όσα είπε. Υπάρχουν αντιφάσεις ε, σε σχέση με τα όσα είπατε. Πρώτον είπατε ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε λέει τίποτα, γιατί είναι τόσο φτωχές οι χώρες. Στη συνέχεια όμω είπατε πρέπει κάτι να κάνουμε εκεί όπου υπάρχει πρόσθετη αξία και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εκεί όπου εμείς εργαζόμαστε όμως μόνο μία πρόσθετη αξία υπάρχει. Μόνο αυτή η πρόσθετη αξία υπάρχει. Δεν υπάρχουν περιτά πράγματα και θέματα ε, που να περιτεύουν λόγω χλειδής. Λοιπόν, Μπορεί να υπάρχει περίοδο περικοπών, αλλά για την παιδεία και εκπαίδευση δεν επιτρέπεται να γίνονται περικοπέ. Αυτά που κάνουμε είναι εξαιρετικά. Το King's Speech το έργο αυτό δεν θα είχε ποτέ τύχει προσοχή αν δεν είχε προαχθεί και δεν είχε βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής ε, όπως έγινε. Να το σκεφτόμαστε αυτό. Πολλά από αυτά που κάνουμε <clears throat> σε σχέση με τα συμφέροντα που υπάρχουν για την παιδεία στα αποπλευράς κρατών μελών όχι μόνο αφορούν αυτά αλλά κάνουμε κάτι που αφορά και τον πολιτισμό, παιδεία, εκπαίδευση, πολιτισμό. Φτάνουμε στο σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη. Ουσιαστικά στις 10 θα έχουμε την έναρξη της ακρόασης. Αν κάποιος δεν έχει κάποια ένσταση μπορούμε να επισπεύσουμε στις 10. Και προτού το κάνω αυτό θέλω να ρωτήσω υπάρχουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις για την συνάντηση των ε, συντονιστών εχθές και τις αποφάσεις σε σχέση με τα πρακτικά για αυτήν δεν υπάρχουν. Εγκρίνονται και επικυρώνονται λοιπόν οι αποφάσεις αυτές ε, τα πρακτικά. Έχει κάποιος αντίρρηση να ξεκινήσουμε τώρα με την ακρόαση. Δεν υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις έτσι. Λοιπόν εντάξει ξεκινάμε τώρα με την ακρόαση για την ε, εκπαίδευση όσον αφορά τα, τους νέους με ειδικές ανάγκες. Disadvantaged youth. Έχουμε προσκαλέσει εξέχουσες προσωπικότητες σε αυτή την εκδήλωση. Την Γιάρμίλα ε, Μπρόσικοφα που είναι ε, δασκάλα σε ένα ειδικό σχολείο κατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης ε, στο σα στην ε, Δημοκρατία της Τσεχίας. Ποια είναι η κυρία αυτή, η κυρία Μπροζίκοβα, παρακαλώ. Βρίσκεται, παρίσταται η κυρία Μπροζίκοβα. Δεν έχει φτάσει ακόμα, έτσι. Βρίσκεται εδώ στην αίθουσα. Ναι. Λοιπόν εντάξει, σας ευχαριστώ. Μετά τη Μαρή Ντόνεραν Γκρίφης που είναι <clears throat> επικεφαλής ε, στην κομιτεία του Δουβλίνου του σώματος που διαχειρίζεται είναι, ε, ε, είναι διευθύνει 22 σχολεία στην κομιτεία του, του Δουβλίνου. Και μετά Χελέν Τερβίν επικεφαλής ε, του σχολείου Weekend School στην Ολλανδία και μετά ο κύριος Μουράτ Μαχντή στο Συμβούλιο α, της ε, Αυστρίας ε, για την Ευρωπαϊκή Νεολαία, Φόρουμ Ευρωπαϊκής Νεολαίας. Θα διακόψουμε για 10 λεπτά, θα τα πούμε στις 10 η ώρα γιατί δεν παρίστανται όλοι. Είναι κατανοητό αυτό γιατί προβλεπόταν για ιστερότερα και όχι για τις 10. Δεν κατηγορώ κανέναν. Α πάρετε ένα καφεδάκι και μετά θα ξανασυναντηθούμε σε 10 λεπτά. Να επανέλθετε όμως, έτσι ευχαριστώ. Cher Πρόεδρος, εντάξει. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ακρόαση για το θέμα ε, παιδεία, εκπαίδευση και παιδιά με ειδικές ανάγκες. Χαιρόμαστε για το ότι η κυρία Βρασικόβα είναι παρούσα από την Τσεχία. Έχουμε την κυρία Γκρίφιν από την Ιρλανδία, Τέρβιν, κυρία Τέρβιν από την Ολλανδία και περιμένουμε και από την Αυστρία τον κύριο Μουράτ Μαχντή από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων. Έχουμε και τον παλαιό νέο μας φίλο Άνταν Ποκόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεφαλής μονάδας για την σχολική εκπαίδευση και το πρόγραμμα Κομμένιους. Αγαπητέ Άνταμ, να θυμάσαι ότι χρειαζόμαστε το πρόγραμμα Κομμένους και μετά το 2013. Αυτό έτσι ως υπενικτική παρατήρηση. Και ξεκινάμε τώρα αυτή την, την ε, ακρόαση. Κάθε μία από εκείνους που θα εκείνες που θα παρέμουν θα, έχουν, θα έχει 10 λεπτά στη διάθεσή της. Θα ακολουθήσουμε και με γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων ανάλογα με το πώς θα συμμετέχουν, ίσως 15 λεπτών. Παρακαλώ επικεντρωθείτε σε ένα συγκεκριμένο θέμα και μην ξεκινήσετε επί παντός του επιστητού να θέτετε ερωτήσεις. Και θα δώσουμε και τον λόγο όπως προτίθεμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να προσθέσω και ένα τεχνικής φύσης σημείο. Αυτή η ακρόαση θα μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Η κάμερα αυτόματα θα στοχεύει στην εισηγήτρια, στην ομιλήτρια που θα ομιλεί εκείνη τη στιγμή. Παρακαλώ όσοι δεν θα παρεμβαίνουν εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα ομιλούν, να σβήνουν τα μικρόφωνά τους, διότι θα παραμένει η κάμερα στραμμένη σε εκείνον που θα έχει το μικρόφωνο αναμένο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτό. Σήμερα το πρωί, χθες, εχθές ήδη συζητήσαμε συχνά για αυτό το θέμα, για τη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση 2020, που ιδιαίτερα τονίζουμε την παιδεία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και την κίνηση των, το κίνημα των νέων, ότι πρέπει να αποφύγουμε να εγκαταλείπουν το σχολείο πρόωρα τόσοι πολλοί μαθητές και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Θα επικεντρωθούμε τώρα σε αυτή την ακρόαση στην ένταξη ε, κοινωνική και σχολική των παιδιών με ειδικέ ανάγκες και για εκείνους που έχουν ε, προβλήματα και φυσικά θα επικεντρωθούμε και στο θέμα εκείνων που πρόωρα εγκαταλείπει το σχολείο. Η κυρία Γιάννη Λαμπρόσικόβα δασκάλα στο, στο σχολείο επαγγελματικής κατάρτισης στο Κρόμεριτς, θα λάβει τον λόγο από την Δημοκρατία τη Τσεχία. Παρακαλώ κυρία Μπρόσικοβα, έχετε τον λόγο. Μεγάλη με τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είμαι καθηγήτρια Ξένες γλώσσες στο κέντρο μαθητείας Κρόμεριτς, στις 400 χιλιόμετρα από την Πράγα. Με ανησυχεί το θέμα των νέων με διανοητική αναπηρία και γι' αυτό και συμμετέχω σε ένα διεθνές ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει στόχο τους ε, νέους ε, διανοητικά ανάπηρους ε, μέσα στο τομέα των ξενοδοχειακών επαγγελμάτων. Το 2005 δε αυτό αποτέλεσε, εντάχθηκε μάλλον απόλυτα στο σχολείο μας. Η ειδική αντιμετώπιση των διανοητικά αναπήρων είναι πρόσφατη. Κατά τη διάρκεια του κομμουνιστικού καθεστώτος ε, οι άνθρωποι αυτοί κρύβονταν γιατί το καθεστώς τους, τους έπιανε και τους ε, φυλάκιζε, τους έκρυβε σε ειδικά κέντρα γιατί θέλαν να δείχνουν ότι το, υπό το σοσιαλιστικό καθεστώς τα πάντα ήταν τέλεια, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Από την ε, μεταρρύθμιση και μετά αρχίσαμε να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, ε, προσπαθήσαμε να γνωστοποιήσουμε τα προβλήματά τους και τις διαφορές τους στον υπόλοιπο πληθυσμό και αυτή τη στιγμή πολλοί κόσμος ε, προσφέρει δωρεές στους ε, διανοητικά ανάπηρους για να <coughs> βελτιωθεί η πρακτική κατάσταση, η υλική κατάστασή τους. Βέβαια, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους δίνουμε τα ψάρια έτοιμα, αλλά να τους μάθουμε να ψαρεύουν το πώς να ψαρεύουν θα το μάθουν μέσα από την πρόσβαση στην κατάρτιση. Ο σχολικός νόμος του 2007 δηλώνει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην κατάρτιση ε, όλοι οι πολίτες, ακόμα και αυτοί που έχουν διανοητικά και σαν απειρίες. η μερική ε, μαθητεία φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική. Εγώ θα περιοριστώ στις δυνατότητες των ατόμων με διανοητικές αναπηρίες να σωματωθούν στα ε, δευτεροβάθμια σχολεία. Σύμφωνα με τις στατιστικές, μόνο 10 με 15% των διανοητικά αναπήρων με λαφριά αναπηρία είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τη βασική εκπαίδευση σε ένα κανονικό σχολείο. Στην ηλικία των 15 ή 17 ετών ένας μαθητής εμάς έχει το δικαίωμα να ε, κάνει την ίδια τάξη δύο φορές μέσα στο πλαίσιο της υποχρεωτικής του εκπαίδευσης όσοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν τη βασική εκπαίδευση έχουν τη, δυνατότητα να παρακολουθήσουν πρακτικό σχολείο για δύο χρόνια όπου μαθαίνουν διάφορα επαγγέλματα, κυπουροί, βοηθοί ε, στα, στα νοσοκομεία, καθαριστές κτλ. για να μπορέσουν να αποκτήσουν το μάξιμο των θεωρητικών γνώσεων. Παραδόξως φαίνεται πως τα επαγγελματικά δευτεροβάθμια λύκεια που προετοιμάζουν τα, παιδιά για διάφορα επαγγέλματα φαίνεται να προσφέρουν δυνατότητες ε, ε, ε, ένταξης και για τα παιδιά αυτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένα άτομο με πνευματική αναπηρία γιατί δεν μπορεί να κάνει τις εξετάσεις, τις εισαγωγικές εξετάσεις. Έχουμε ένα πρόγραμμα που συμμετέχουμε σε στην ανάπτυξη σχολικών προγραμμάτων για τρία χρόνια με τίτλο «Ρεστό du Antiquaire» Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της ε, Φλωρεντίας στην Ιταλία ε, που έχει μεγάλη εμπειρία με, του, για, για τα άτομα με διανοητικές αναπηρίες το σχολείο μας συμμετέχει και στόχος είναι να διευκολυνθεί η αυτονομία των ε, τρισομικών νέων χάρη στην ένταξή τους ε, στην ε, κατάρτιση στη ξενοδοχειακά επαγγέλματα και μέσω της πρόσβασής τους στον κόσμο της εργασίας. Γιατί τα παιδιά με σύνδρομο Down, γιατί ενδιαφέρονται για αυτόν τον ε, επαγγελματικό κλάδο, είναι πιο εύκολο, δεν χρειάζεται συγκεκριμένες δεξιότητες ή συγκεκριμένες τεχνικές. Αντίθετα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα που έχουν για εύκολη επαφή με τους άλλους. Είναι πολύ επικοινωνιακή, χαρούμενη, χαρμογελαστή και εξυπηρετική, ειδικά ε, καλή στη εστιατόρια. Επιπλέον, τα παιδιά με σύνδρομο Down ζουν αυτή τη στιγμή περισσότερο χρονικό διάστημα χάρη στις πρόοδους της ε, ιατρικής και οι γονείς τους δεν μπορούν να βρίσκονται πάντα στο πλάι τους. Εμείς πήγαμε στο κέντρο, το ειδικό κέντρο της πόλης μας, όπου ε, πήραμε ένα τρισομικό παιδί, το οποίο ε, παρακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα πιλωτικό μαζί με τους εκπαιδευτές μας. Ε, πρόκειται για ένα πείραμα και γι' αυτό μας επιτράπηκε να το φιλοξενήσουμε μέσα στις εγκαταστάσεις μας. Αυτός ο νέος πειραματικός μαθητής μας καταρτίστηκε για τρία χρόνια στα επαγγέλματα των εστιατορίων παρακολουθήθηκε από τους ε, δικούς μας καθηγητές και την τρίτο χρόνο έκανε και ένα στάζ σε ένα εστιατόριο όπου οι πελάτες πολύ σύντομα συνήθισαν ε, την παρουσία του και το αφοπλιστικό του χαμόγελο μάλιστα ε, προσέλκυσε και νέους πελάτες, κυρίως νέους. Αυτά τα παιδιά, αυτό το παιδί έκανε φοβερές προόδους, μπόρεσε να χειριστεί ακόμα και την προετοιμασία κοκτέιλ και κυρίως έχει ε, κυρίως μέσω της μίμησης ε, της συμπεριφοράς των ε, συναδέλφων του. Δεν κοιτά πια τους άλλους με ανοιχτό το στόμα, δεν σέρνει τα πόδια του. Επίσης παρακολούθησε θεωρητικά μαθήματα αγγλικών, πληροφορικής και μπόρεσε να συντάξει και ένα σύντομο μενού στον υπολογιστή. Πήγε και σε στάζ στη Γαλλία και στην Ιταλία η παρουσία του είχε τεράστιο αντίκτυπο δε στους συμμαθητές του, καθώς και στο προσωπικό του σχολείου μας. Οι μαθητές των άλλων τάξεων τον ζητούσαν για τα πρακτικά μαθήματα, όλοι προσπαθούσαν να τον εθαρρύνουν και να μοιραστούν μαζί του τη χαρά του. Και α, εκείνος μας έμαθε να είμαστε πιο ευαίσθητοι και ε, ξύπνησε την ανθρωπιά μας. Τα τρία ευρωπαϊκά σχολεία θέλησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία μέσω των προγραμμάτων μας. Όμω, το τελικά δεν έγινε δεκτή η πρόταση. Το παιδί αυτό επανήλθε στο Ίδρυμα ε, α, δυστυχισμένο, η υγεία του επιδεινώθηκε και ξαναβρήκε τις κακές του συνήθειες. Ελπίζαμε να πετύχουμε κάποιο συμβόλαιο, κάποια σύμβαση εργασίας σε κάποια επιχείρηση. Ε, χωρίς όμως ε, προστατευμένη ε, ε, εργασία. Χρειάζεται ωστόσο νομική κάλυψη για την υπογραφή της Σύμβασης Εργασίας Το Έγιναν διαβήματα ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης και στο Υπουργείο Εργασίας. Τελικά δεν κατέληξαν όμως πουθενά. Ε, υπήρξε, υπήρξαν πάντα ίδια ίδιοι δισταγμοί και αντιρρήσεις. Ο καθηγητής του το επέτρεψε να επανέλθει στο σχολείο ώστε τουλάχιστον να παρατηρεί τους συμμαθητές του οι οποίοι είχαν περισσότερη τύχη στη ζωή ο δε ο επιθεωρητής μας, διευθυντής αποφάσισε να προβεί σε δράσεις ε, με δική του ευθύνη και επέτρεψε στο παιδί αυτό να επανέλθει στο σχολείο για κάποιες, κάποια προπαρασκευαστικά μαθήματα και να συμμετέχει στις διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις όπου οι μαθητές της σχολείου μας προσφέρουν ε, γεύματα ή αναψυκτικά. Ελπίζουμε λοιπόν πως θα μπορέσουμε ε, να βρούμε με αυτόν τον τρόπο το μελλοντικό του εργοδότη. Κάναμε και μια μικρή δημοσιο... δώσαμε κάποια δημοσιότητα στο τοπικό τύπο. Ορισμένοι συνειδητοποίησαν ότι δώσαμε κάποιες ευκαιρίες και λόγο στους διανοητικά ανάπηρους Ελπίδα μας ε, είναι μια ημέρα των υπερών να μπορέσουμε να δώσουμε θετικές απαντήσεις στις οικογένειες των παιδιών με διανοητικές αναπηρίες και να ε, ε, μπορέσουμε να δώσουμε στο σχολείο μας ένα κεντρικό ρόλο για την ένταξη ε, των παιδιών αυτών στις δομές κατάρτισης αλλά και να παίξουμε διάμεσο ρόλο με τις επιχειρήσεις και να τους διοχετεύσουμε στους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα εκπροσωπηθούν από κάποιον ε, νομικό εκπρόσωπο για τη συμπογραφή των συμβάσεων εργασίας και να μην χρειαστεί να επανέλθουν στα ειδικά σχολεία, να έρθουν στα επαγγελματικά λύκη και να εξασφαλίσουν και την διαβίου κατάρτισή τους. Έτσι καλούμε και τα άλλα ε, ξενοδοχειακά σχολεία να παρακολουθήσουν το παράδειγμά μας, ε, προτείνουμε την βοήθειά μας με τη βάση της εμπειρίας μας. Όλοι γνωρίζουμε καλά ότι οι διανοητικά ανάπηροι δεν θα συμβάλλουν ποτέ στην οικονομική ευημερία της χώρας τους. Έχουν όμως ε, τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους γιατί μας μαθαίνουν να σεβόμαστε την διαφορετικότητα του άλλου και να σεβαστούμε την διαφορά του άλλου οδηγεί στην ανεκτικότητα και η ανεκτικότητα καθιστά τον κόσμο μας λιγότερο επικίνδυνο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Μπροσικόβα. Θα παρακαλέσω τους Τσέχους συναδέλφους να ασχοληθούν λίγο με το δικό σας πρόβλημα. Κυρίως πρέπει να ασκήσετε πιέσεις στους Τσέχους εθνικούς βουλευτές, αλλά και τους ευρωβουλευτές. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα μιλήσω με τους Τσέχους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο, τους ευρωβουλευτές, να ασχοληθούμε με αυτή την πλατφόρμα στη χώρα σας για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα, γιατί είναι τεχνικό το πρόβλημα. Βέβαια, πρώτα πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες και μετά τα υπόλοιπα. Ζητώ συγγνώμη, εγώ φταίω, θα τα συζητήσουμε μετά. Η κυρία Μαρή Ντόνελαν Γκρίφιν. Good morning. Καλή σας μέρα. Είμαι Διευθύντρια Επικεφαλής ε, της Κομιτείας ε, Δουβλίνου Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάτησης. Ε, σε σχέση με τον επαγγελματικό τομέα στην Ιρλανδία παρέχεται το ίδιο φάσμα μαθημάτων όπως και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε 26 σχολεία τα οποία έχουμε υπό την δική μας εποπτεία έχουμε κινηθεί και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε ακριβώς με την... Ε, πιο αργά. Ε, ε, λέτε. Εντάξει. Να επιβραδύνουμε λίγο. Επειδή ήμουνα δασκάλα και είχα συνηθίσει να μιλάω πιο γρήγορα, εν πάση περιπτώσει, στην κομιτεία του Δουβλίνου η Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει αυτά τα σχολεία υπό την εποπτεία της ήμουν επικεφαλής σε ε, ειδικό σχολείο με ε, άτομα με ειδικές ε, ανάγκες και για άλλους μαθητές. Τοποθετούμε λοιπόν σε σχέση με τους νέους με ειδικέ ανάγκες στην Ιρλανδία υπό το, τη δική μου πείρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών στόχων στην ε, Λισαβόνα, στην ε, ημερήσια διάταξη της Σαβόνας, ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης και της παιδείας και η κοινωνική ένταξη η ανάπτυξη ε, εκπαιδευτικών συστημάτων που να είναι κοινωνικά να βοηθούν στην ένταξη είναι ένας από τους κύριους στόχους όσο έχουμε τέτοια σχολεία για την ένταξη στην ε, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με λιγότερες διαφορές ε, σε σχέση με μαθητές, ε, μικρότερη διακριτική μεταχείριση όσον αφορά διαφορετικής προέλευσης μαθητές. Έχουμε το δευτεροβάθμιο επίπεδο στην Ιρλανδία που έχει αναπτυχθεί προς τον 21ο αιώνα και λαμβάνοντας υπόψη τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα οι ευκαιρίες που δίνονται σε σχέση με τις δυνατότητες αυτές είναι υψηλέ. Σε σχέση με τη δεκαετία του 90 πέτυχε η Ιρλανδία ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανάπτυξη παγκόσμια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει υψηλό ποσοστό επιστροφή ε, όσον αφορά του νέου αυτού ε, στην ε, αγορά εργασία. Οι εξελίξει σε αυτή την περίοδο δείχνουν ότι η οικονομική ανάπτυξη αφεαυτής ε, δεν μπορεί να εκριζώσει την φτώχεια ή τις κοινωνικές ανισότητες. Η Ιρλανδία έχει σχετικά υψηλά ποσοστά ανισότητας ε, που αντανακλώνται και σε σχέση και με την ε, κατοικία και την, την δυνατότητα διαβίωσης των πολιτών. Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό σε σχολεία και αυτό έχει πολλαπλασιαστικό, πολλαπλασιαστική επίπτωση θα μπορούν οι γονείς να επιλέγουν τα σχολεία στα οποία στέλνουν ε, τα παιδιά τους και πραγματικά ε, παίρνουν η δυνατότητα επιλογής ε, τοπικών σχολείων, ιδιαίτερα για την μεσαία τάξη, δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση σε σχέση με τον ανταγωνισμό ε, όσον αφορά τις ε, ε, διάφορες θρησκευτικέ ομολογίες υπήρχε ένα συγκεκριμένο ποσοστό έναντι της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ενώ ο τομέας της επαγγελματικής κατάρτισης είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας, οι επιπτώσεις αυτού του κατακαιρματισμού είναι σημαντικές, ιδιαίτερα οι επιπτώσεις εις βάρος των παιδιών με μειονεξίες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Υπήρχε μια, υπήρξε μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το πλαίσιο για την εκπαίδευση ατόμων με ειδικέ ανάγκες στην Ιρλανδία από τα τέλη του 1990. Το 1998 ε, καθορίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόσβαση σε τέτοιο σχολείο για οποιοδήποτε άτομο έχει ανάγκη τέτοια ειδική εκπαίδευση, ε, λαμβάνοντα πάντα υπόψη τι ειδικέ ανάγκε που υπάρχουν για τέτοιου μαθητέ. Ε. Αυτό σε σχέση με την παιδεία εκπαίδευση για άτομα με ειδικέ ανάγκε που ολοκληρώθηκε ολοκληρώθηκε μέχρι το 2005. Τα τρία αυτά νομοθετήματα καθορίζουν τις υποχρεώσεις ε, από πλευρά των φορέων ε, προς ε, τους μαθητές με ειδικέ ανάγκες βλέπουμε ότι σε σχέση με τα κονδύλια υπάρχουν συγκεκριμένες επιπτώσεις και όπως όλοι γνωρίζουν υπάρχουν πολύ λιγότερα κονδύλια σήμερα στην Ιρλανδία διαθέσιμα από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Παρ' αυτά όμως υπήρξε σημαντική αύξηση του αριθμού των παιδιών με ειδικέ ανάγκες και η πολιτική ένταξη παιδιών με ειδικέ ανάγκες είναι κάτι το προφανές ως ανάγκη που πρέπει να ε, αντιμετωπίζεται. Σε σχέση με την ε, Τσεχία όπου οποιαδήποτε παιδιά με ανάγκη με ειδικές ανάγκες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια σχολεία. Ε, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση και η κατάρτιση, οι δεξιότητες, οι ικανότητες όποτε ε, πρέπει, πρέπει να προσφέρονται. Ενώ τα περισσότερα σχολεία, δευτεροβάθμια σχολεία έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση τα άτομα με ειδικέ ανάγκες σε αυτά. Δεν φεύγουν πάντα με διπλώματα ή πτυχία από αυτά οι μαθητές. Να επιβραδύνω ναι, και από την νοτιοδυτική Ιρλανδία. Διαβάζεται υπερβολικά γοργά. Εσείς δεν, δεν έχει σχέση με το από πού προέρχεστε. Διαβάζετε πάρα πολύ γρήγορα. Παρακαλώ να επιβραδύνετε λίγο το ρυθμό σας. Προέρχομαι. Δεν χρειάζεται να τα διαβάσετε όλα. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, κάποια ιδέα να μας την εκθέσετε σε αδρές γραμμές. Έρχομαι από το Κέρι όπου μιλάμε πολύ γρήγορα. Τι να κάνω. Η δυσκολία βρίσκεται με τα παιδιά με ειδικέ ανάγκε, δεν μπορούν να πάρουν πάντα ένα πτυχίο και δεν ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και έτσι δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπως όλοι οι άλλοι ε, μαθητές. Το 2008 και αυτό αναφέρεται σε αυτό το οποίο ανέφερα προηγούμενα για την ε, την επίπτωση πολλαπλασιαστή. Συντάχθηκε μία μελέτη και βρέθηκε ότι σε κάποια σχολεία, και πάλι εδώ κάνω λόγο για τον επαγγελματικό τομέα, τομέα επαγγελματικής κατάτησης, ότι έπαιρναν πολλού, πολλούς περισσότερους μαθητές με ειδικέ ανάγκες από ότι άλλα σχολεία. Και αυτό συνεχίζει να είναι ένα χαρακτηριστικό Υπάρχει και η αναγνωρισμένη ανάγκη να υπάρξει καλύτερο συντονισμό σε σχέση με τι υπηρεσίε στο κρατικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και επειδή υπήρξαν τόσε πολλέ αλλαγέ όσον αφορά την νομοθεσία κατά τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα, δεν υπήρξε επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουμε το σχολικό σύστημα για την απορρόφηση των μαθητών με ειδικέ ανάγκε. Δεν έχει καταρτιστεί το εκπαιδευτικό προσωπικό ακόμα όπω πρέπει και υπάρχει μικρή υποστήριξη για τα παιδιά με ειδικέ ανάγκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια δυσκολία ξεχωριστή είναι το ότι τα σχολεία ενώ λειτουργούν με στόχους ε, ένταξης δεν προχωρούν σε αυτή την ολοκλήρωση. Γιατί αυτό θα σήμερα θα έπρεπε να αλλάξουν ε, οι ε, διεργασίες και πολιτικές ε, για την ένταξη των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Σε μια περίοδο συγκυρίας, οικονομικής συγκυρίας λιτότητας και περικοπών, περικόπτουν τα κονδύλια και τα άτομα με ειδικέ ανάγκες αντιμετωπίζουν μεγάλη, μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τη σχολική τους εκπαίδευση. Υπάρχει και το θέμα της ανισότητας ε, και της μη επαρκούς επίδοσης. Ε, εδώ τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες απαιτούν ε, ειδική υποστήριξη και ειδικά προγράμματα για να μπορέσουν να αντισταθμιστούν αυτές οι ανισότητες στην Ιρλανδία δεν καταφέρνουν από την ε, πρωτοβάθμια να περάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών και εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να έχουν κάποια ε, διπλώματα. Έχουν και δυσκολίες ε, στο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα δυσλεξίας και να μάθουν και καλά να διαβάζουν και να γράφουν. Και προσπαθούμε να ε, στοχοθετήσουμε αυτές ε, τις ε, ανάγκες. Χρειάζονται ιδιαίτερες, ιδιαίτερα κονδύλια ώστε να μάθουν να διαβάζουν, να κάνουν αριθμητικούς υπολογισμούς. Υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης και από τους γονείς. Συνεργάζονται τα σχολεία και με άλλους φορείς για να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Και ζητήθηκε πρόσφατα από τα σχολεία να ε, στοχοθετήσουν ε, με συγκεκριμένα προγράμματα αυτές τις ανάγκες και η εποπτεία, η επιθεώρηση εκπαίδευσης ε, ελέγχει το τι γίνεται. Όμως υπάρχουν και ανισότητες εις βάρος των μαθητών πολλές φορές. Αυτές οι πρακτικές με αργούς ρυθμούς αντιμετωπίζονται και από την επιθεώρηση εκπαίδευσης και βλέπουμε ότι μετά τον ε, ε, καθορισμό των ε, κέντρων νεότητας για την κατάρτιση των νέων πάνω από τα 16 υπάρχει ανάγκη να επικεντρωθούμε στην μειονότητα ε, της ηλικίας κάτω από 16, ιδιαίτερα για τα αγόρια που έχουν προβλήματα και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και με το νέο Υπουργείο στην Ιρλανδία για τα παιδιά και την παροχή υπηρεσιών στα παιδιά θα αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Έχουμε την, ε, το στόχο ώστε να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το ε, θέμα της ε, ε, ολοκλήρωσης της, του κύκλου σπουδών με υψηλό βαθμό, ωστόσο δεν υπάρχουν θέσεις απασχόλησης στην αγορά εργασίας και αυτό είναι αρνητικό. Καλωσορίζουμε την δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης των παιδιών γιατί όσο περισσότερες ικανότητες αποκτούν τόσο περισσότερες προοπτικές έχουν να απασχοληθούν βρισκόμαστε σε ένα χαμηλότερο ποσοστό, σε 73% και πάλι ε, τα αγόρια έχουν ένα ε, χαμηλότερο ποσοστό από ότι τα κορίτσια και βλέπουμε εδώ την ανισότητα και σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Είναι απόδειξη για ε, την πρόσθετη αξία που παρέχεται από τα πρόσθετα κονδύλια που δίνονται στα σχολεία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Όμως οι φτωχότεροι ε, μαθητές σε σχέση με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγώ ίδια είχα εμπλακεί σε ένα πρόγραμμα που προσπαθούσε από περιοχές με προβλήματα να βοηθήσει ε, άτομα να περάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλή δουλειά πρέπει να γίνει όμως ακόμα για αυτή την ένταξη. Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ιρλανδία εξακολουθεί να ε, στεγανοποιείται όσον αφορά την διαφορά των φύλων. Υπάρχουν πολλά σχολεία τα οποία είναι αποκλειστικά σχολεία μόνο για αγόρια ή για κορίτσια. Υπάρχει η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πιο ευάλωτων. Ε, υπάρχουν κενά που πρέπει να καλυφθούν. Υπάρχει ανάγκη να προβληματιστούμε και να καταρτήσουμε μια κοινή πολιτική για αυτά τα θέματα παιδείας και πρέπει να δούμε και την παροχή υπηρεσιών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Περισσότερα αγόρια, ιδιαίτερα από περιοχές με μειονεξίες, φτωχότερες ε, περιοχές ε, βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μια σημαντική αύξηση των ποσοστών συμμετοχής δεν σημαίνει υποχρεωτικά πρόοδο που επιτυγχάνεται στην άση των ανισοτήτων. Ακόμα και σε μαθήματα μετά το σχολείο βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές ε, όσον αφορά τις επιδόσεις των μαθητών ανάλογα με την προέλευσή τους. Πρέπει να δούμε τη δημιουργία οικονομικών προϋποθέσεων ε, για μεγαλύτερη ε, ευημερία και ανάπτυξη και μεγαλύτερη συμμετοχή. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να μεγαλώνει αυτό το χάσμα εκείνων που αποκλείονται από τη γνώση και περιθωριοποιούνται. Και στην Ιρλανδία έχουμε έναν μικρό αριθμό ε, πολύ περιθωριακών ατόμων που λόγω αυτής της κατάστασης επιδεινώνεται η, κατάσταση στην οποία βρίσκονται ως περιθωριοποιημένα άτομα. Πρέπει να κάνουμε να επανορθώσουμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Τώρα κύριε... λόγο, Τερβέιν, παρακαλώ. Ονομάζομαι Ελένη Τερβέιν. Έχω ιδρύσει ε, το σχολείο του ε, Σαββατοκύριακου. Είναι κάτι σαν φροντιστήριο για το Σαββατοκύριακο για μειονεκτικέ συνοικίες στην Ολλανδία. Μου ζήτησαν να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα, με χαρά να το κάνω. Για να σας δώσω ε, μια ε, εικόνα για την εκπαίδευση, να είναι μια εκπαίδευση πιο ελκυστική, πιο συμπληρωμένη, πιο ολοκληρωμένη. Έχω ένα δεκάλεπτο ε, για να σας εξηγήσω πώς είναι αυτό το σχολείο, πώς μας υποστηρίζει η κοινωνία των πολιτών, τι παρέχουμε και τι σχέδια έχουμε για το μέλλον και πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένω να συνεργαστούμε μαζί σας. Τι είναι το σχολείο, σας είπα, είναι συμπληρωματικό, είναι φροντιστήριο. Τρία χρόνια κάθε Κυριακή ε, μέχρι ηλικίας 14 ετών ε, και ε, έρχονται διάφοροι ειδικοί εμπειρογνώμονες, δημοσιογράφοι, γιατροί, δικηγόροι, από όλα τα επαγγέλματα, καλλιτέχνες που εξηγούν το επάγγελμά τους αλλά συνεργάζονται και με τα παιδιά. Οι δημοσιογράφοι ας πούμε ε, κάνουν και πρόγραμμα ή εφημερίδα. Οι γιατροί μαζί με τα παιδιά. Βεβαίως δεν θα κάνουν εγχειρήσει με τα παιδιά, αλλά κάνουν πολλά άλλα πράγματα σε συνεργασία με τους μαθητές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει έρθει και έχει διδάξει και επίσης οι απόφοιτοί μας έρχονται μια φορά το χρόνο στις Βρυξέλλες και κοιτούν πώς δουλεύουν οι ευρωπαϊκοί θεσμικά όργανα. Αυτό το σχολείο λοιπόν του Σαββατοκύριακου ε, υπάρχει ε, τα τελευταία 13 χρόνια. Έχουν έρθει 2.000 ε, επαγγελματίες εθελοντικά, δεν πληρώνονται και έχουμε πάντα κόσμο. Δεν είχαμε ποτέ δυσκολία να βρούμε εθελοντές να έρθουν να διδάξουν. Ε, γιατί θέλουν να βοηθήσουν και είναι τεράστια η συμβολή αυτή για παιδιά του γυμνασίου από μειονεκτικέ συνοικίε. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα να βρούμε καθηγητέ και είναι πολύ μεγάλη υποστήριξη τη κοινωνία των πολιτών και μάλιστα μα ε, ε, χρηματοδοτούν. Ε, γιατί δεν μας χρηματοδοτεί το κράτος, αλλά ιδιώτες. Εννέα τέτοια σχολεία υπάρχουν σε όλη την Ολλανδία από 2,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ο προπολογισμό που πρέπει για να τον βρούμε, να αγωνιστούμε σκληρά, αλλά τον βρίσκουμε από ιδρύματα, από εταιρείε και ε, πραγματικά ξέρουν, καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι αυτοί ότι η επένδυση ε, στο μέλλον περνάει μέσα από την επένδυση στην παιδεία και στην κοινωνία και το καταλαβαίνουν. Και ακριβώς ε, για νέους ε, που έχουν ενδεχομένω και κάποιε ειδικέ ανάγκε ή διανοητική αναπηρία χρειάζεται η κοινωνία και μπορεί να υποφελείται και από του ίδιου η κοινωνία. Τι κάνει το σχολείο μας. Μπορείτε να το δείτε αυτό με το καλύτερο τρόπο από τους αποφύτου μας. Σας είπα ότι 13 ε, χρόνια έχουμε κάνει αυτή την προσπάθεια. Ε, οι μαθητές που άρχισαν την πρώτη χρονιά 10 ετών είναι τώρα 23. Και έρχονται και πρώην μαθητές μας, απόφοιτοι, και κάνουν μάθημα. Ε, κάνουν σπουδές τώρα. Και αυτό λέει και το σχολείο του Σαββατοκύριακου. Τους λέμε... Στο κανονικό σχολείο, το καθημερινό, ε, σας υποχρεώ να πάρετε πτυχίο. Μόνο το ΝΑΤΟ το πτυχίο θεωρείται επιτυχία. Στο δικό μας σχολείο αξιοποιείται η δυνατότητα και η αξιότητα και ε, η δεξιότητα κάθε μαθητού. Και αν ε, συγκρίνουμε κάποιες ομάδες μαθητών, γιατί έχουν γίνει και τέτοιες μελέτες, με, με μια ομάδα μάρτυρα, ας πούμε, από το κανονικό σχολείο και από το δικό μας σχολείο, οι δικοί μας μαθητές είναι πολύ πιο ενθουσιώδεις, είναι πολύ πιο ε, επιμελείς, ε, προσιλωμένοι και έχουν και κίνητρα να συνεχίσουν. Και θέλουν να επενδύσουν και μαθαίνουν να επενδύουν και στον εαυτό τους και στην κοινωνία. Και μετά έρχονται και κάνουν μάθημα στους καινούριους μαθητές. Ε, τα σχέδια για το μέλλον δεν είναι να εξαπλωθούμε σε όλη την Ολλανδία, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον τρίτο κόσμο για διάφορους λόγους μεταξύ αυτών ε, και οικονομική, αλλά εγώ πιστεύω ότι ε, θα πρέπει και μπορεί να αναμειχθεί πολύ περισσότερο η κοινωνία των πολιτών στο κανονικό σχολείο, εκτός από το σχολείο του Σαββατοκυριακού. Γι' αυτό δεν θέλουμε να επεκταθούμε. Θέλουμε αυτή η προσπάθεια να ε, διοχετευτεί και προς το κανονικό σχολείο. Ε, υπάρχει αρκετός χώρος. Λοιπόν, η δική μας αποστολή στην Ολλανδία πλέον είναι να περάσουμε ε, ε, σε μεγαλύτερη ενσωμάτωση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διεθνώς θα μας ενδιαφέρε όμως να ιδρύσουμε και τέτοια σχολεία προσεχώς στο Βερολίνο, στο Παρίσι, γιατί όχι και στις Βρυξέλλες, για να μεταφέρουμε και διεθνώς την εμπειρία μας αυτή. Επίσης, κάποιες πρωτοβουλίες ε, που έχουμε εμπνεύσει να ε, συνεχιστούν και ακούω ότι η Μαρή που είναι ευρωβολευτής των Φιλελευθέρων προγραμματίζει ένα ευρωπαϊκό θερινό πανεπιστήμιο European Summer School και μας έχει ζητήσει και την υποστήριξή μας για να γίνει αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή ένα αντίστοιχο πρόγραμμα αυτό που κάνουμε εμείς σε μαθητές του γυμνασίου από τα διάφορα κράτη της Ευρώπης με ανταλλαγές ε, το καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια αυτή και πολύ αξιόλογη. Τι θέλουμε λοιπόν να κάνουμε εμείς στο μέλλον. Να τονίσουμε ότι Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, ε, του φροντιστηρίου το Σαββατοκύριακο ε, από την κοινωνία με επαφή με επαγγελματίες, με καλλιτέχνες όπως είπα επιστήμονες. Είναι πάρα πολύ σημαντική για τα παιδιά του γυμνασίου και θα πρέπει να συνεχιστεί και να επεκταθεί και στην κανονική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά να δείξουμε και στην Ευρώπη ότι είναι σημαντικό η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει και ε, να έχει επαφή με μαθητές του γυμνασίου που από την κοινωνική τους προέλευση και καταγωγή δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να έρχονται σε επαφή με αυτούς τους κλάδους κοινωνίας. Και στόχος είναι να προετοιμάζονται οι νέοι μαθητές για να διαδραματίζουν ένα πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Και όταν μιλάμε με νέου, ή ασχολούμαστε με του νέου, να μην κοιτάμε πάντα τι πάει στραβά με του ε, νέου ή με του εφήβους, αλλά από την ηλικία των 10 ετών να τους ε, παίρνουμε από το χέρι, να του συνοδεύουμε, να του βοηθούμε για να του προετοιμάζουμε να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών. Γι' αυτό η επένδυση στον ενθουσιασμό, στην όρεξη για μάθηση είναι η λέξη κλειδί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και με στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τερβάιν. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Μουράτ Μαχίδη, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φόρουμ των Ευρωπαίων Νέων. Θα είμαι ε, σύντομος και θα μιλήσω στα αγγλικά, γιατί συνήθως ε, μιλάω αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε να σας παρουσιάσω τις απόψεις του φόρου μας εδώ για θέματα που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Για όσους δεν μας γνωρίζουν, το Φόρουμ των Ευρωπαίων Νέων είναι ένα εξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί πάνω από 100 εθνικές οργανώσεις νέων και συμβούλια νέων από όλη την Ευρώπη. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους νέους να συμμετέχουν ενεργά στην Ευρώπη, ε, στην κοινωνία, να βελτιώσουν τη ζωή... Ε, Κοιτάξτε, εσείς Ιρλανδός δεν είστε. Μπορείτε να μιλάτε πιο αργά, λέει η πρόεδρος. Slower, slower. Και μπορείτε να διαβάζετε ε, ε, πιο αργά ή ακόμα καλύτερα να μιλάτε, που έτσι και αλλιώς θα μιλάτε πιο αργά youth. Λοιπόν, μιλούμε για ε, τους νέους σε μειονεκτική θέση, μαθητές σε μειονεκτική θέση. Ε, θα πρέπει η κοινωνία να επιτρέπει σε όλους να αναπτύξουν την προσωπικότητα και την ικανότητά τους. Αυτό σημαίνει ε, ισχυρά μέτρα πολιτικής και ε, ένα ισότιμο σύστημα με ίσες ευκαιρίες για την εκπαίδευση. Δυστυχώς ε, παραμένει ε, μεγάλη η σύνδεση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των γονέων με ε, την εκπαίδευση των νέων. Αυτό θα πρέπει να σπάσει, έτσι ώστε οι νέοι που έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αναπτυχθούν και αυτοί πλήρως. Πάντα τονίζουμε τη σημασία των δικαιωμάτων, αλλά μέσα στα δικαιώματα είναι το δικαίωμα στην εκπαίδευση και αυτό αναγνωρίζεται από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο οι νέοι δεν θα πρέπει να θεωρούνται μόνο κάτοχοι δικαιωμάτων, δικαιούχοι, αλλά θα πρέπει να θεωρούνται και κάτοχοι και ιδιοκτήτε τη ίδια τη εκπαίδευση, να αποφασίζουν εκείνοι ε, τι θα επιλέξουν ω δρόμο μονοπάτι για την εκπαίδευσή του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και οι νέοι μαθητέ να ε, αποφασίζουν με τα λόγου γνώσεω για το πότε θα σταματάει η εκπαίδευσή του πότε θα ολοκληρώνεται και βάση με τα σχέδια για την καριέρα τους και τις προσωπικές αποφάσεις. Δηλαδή η ε, πρόορη εγκατάλειψη ε, του ε, σχολείου μπορεί να είναι προσωρινή, δεν είναι ανάγκη να είναι οριστική. Μπορεί κάποιος να αλλάξει η γνώμη, να αρχίσει μια νέα εκπαιδευτική πορεία. Τι βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη. Το βασικότερο στοιχείο για το εάν εγκαταλείπει πρόωρα ένα παιδί το σχολείο είναι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της οικογένειάς του. Δεν είναι πάντα ίσες ευκαιρίες ε, από πλευράς πολιτιστικού ή ανθρώπινου κεφαλαίου η υποστήριξη της οικογένειας. Επίσης, ε, τα σχολεία ε, μεταβιβάζουν γνώση χήμα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να ε, μαθαίνουν ε, κάποια πράγματα παιδιά, αλλά όχι κάθε παιδί ξεχωριστά ε, σύμφωνα με τις δεξιότητες και τις ικανότητες του. Και τελικά έχουμε κοινωνικές ανισότητες και πρόλη εγκατάλειψη του σχολείου. Το μακροχρόνιο κόστος και το οικονομικό και το κοινωνικό είναι πολύ μεγάλο και για την κοινωνία και για τους νέους τους ίδιους. Πολλέ από τις ανεπιθύμητε συνέπειε της πρώτη εγκατάλειψη σχολείου ε, συνδέονται ε, μεταξύ τους και δημιουργούν ένα ε, φαύλο κύκλο και τελικά αποκλεισμό των νέων αυτών. Μεγαλύτερη φτώχεια, Μάλλον η φτώχεια οδηγεί σε μεγαλύτερο κίνδυνο να διακόψει κανεί νωρίτερα το σχολείο, άρα και σε ακόμα μεγαλύτερη φτώχεια. Τώρα, τι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό. Το ε, καλύτερο επίπεδο είναι το σχολείο και η κοινότητα, όσο γίνεται πιο κοντά στο μαθητή. Σε τοπικό επίπεδο και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν όμω και εθνικέ και ε, ευρωπαϊκέ πολιτικέ. και θα πρέπει να είναι και εγκάρσιες αυτές οι πολιτικές. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη δεδηλωμένη πρόθεση και δέσμευση για ε, ε, την ατζέντα για νέε δεξιότητε και ε, θέσει απασχόληση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν αργεί αυτό. Θα πρέπει τα διάφορα εμπόδια κοινωνικά και οικονομικά που εμποδίζουν του νέου να φτάσουν στην ανώτατη και ανώτερη εκπαίδευση να αρθούν. Κανείς να μην μένει πίσω παρά τη θέλησή του. Και θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία στο ανθρώπινο, στο οικονομικό δυναμικό έτσι ώστε τα συστήματα αυτά τα εκπαιδευτικά να εκπαιδεύουν όλο τον κόσμο χωρίς ε, διακρίσεις και να μην απευθύνονται αποκλειστικά σε ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Τα προγράμματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και στο κέντρο του εκπαιδευτικού συστήματος να είναι ο μαθητής Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες ανάγκες των νέων με σωστά πτυχία και διπλώματα έτσι ώστε ε, ο κάθε μαθητής να έχει ένα ενδεικτικό, να έχει ένα πιστοποιητικό, ένα δίπλωμα που να αναφέρει τα ε, προσόντα τις δεξιότητες και ικανότητες που έχουν, χωρίς να είναι το ανώτατο δίπλωμα του σχολείου. Ε, για να μπορεί να αποδεικνύει ο μαθητής, ε, αν θέλει στη συνέχεια να ε, συνεχίσει τις σπουδές του, μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει. Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθούν τα προγράμματα για τους νέους να έχουν δυνατότητες εναλλακτικής εκπαίδευσης μαθητείας και μη ακαδημαϊκές δεξιότητες. Θα πρέπει ε, όμως να γίνουν όλα αυτά ε, με τρόπο αυτόνομο, να διαλέγουν οι μαθητές οι ίδιοι τι θέλουν, χωρίς εξωτερική πίεση. Αυτό είναι κάτι που λείπει ε, σήμερα στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Επαναλαμβάνω, δεν είναι θέμα οικονομικό. Και εγώ, είναι θέμα δικαιωμάτων, εκπροσωπώ ε, ένα φόρουμ ε, οργανώσεων νέων και θέλω να τονίσω και τα θετικά αποτελέσματα και το θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανώσεις των νέων ε, για την καταπολέμηση και πρόληψη της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. Υπάρχει και η άτυπη εκπαίδευση προς τους νέους και στις οργανώσεις νέων. Έτσι αυξάνεται η αυτοπεποίθηση, τονώνεται ο αυτοσεβασμός και οι ε, κοινωνικές δεξιότητες και πέφτουν οι φραγμοί ε, που υπάρχουν ε, στο κλασικό σχολείο και στην αγορά εργασίας. Και επίση έρχονται να καλύψουν οι οργανώσει των νέων τα κενά που αφήνει η εκπαίδευση και φέρνουν στα σχολεία ε, και το σύστημα της άτυπης εκπαίδευσης είναι στο κέντρο ο μαθητής και το σχολείο γίνεται πιο ελκυστικό. Συμμετέχουν περισσότερο οι νέοι ε, στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, ε, φοιτητικοί σύλλογοι σε σχολεία μπορούν να εξηγήσουν στους μαθητές του γυμνασίου πώς θα έχει η ζωή τους αργότερα, να έχουν τη δυνατότητα επιλογής ε, οι μαθητές πότε θα φύγουν από το σχολείο και ε, βέβαια δεν μπορούμε εμείς ή η άτυπη εκπαίδευση να διορθώσουμε τα στρεβλά της επίσημης εκπαίδευσης. Μπορούν όμως τα σχολεία έτσι να καταλάβουν περισσότερο τις ανάγκες των μαθητών, τις προσδοκίες των μαθητών ε, και ιδιαίτερα των μαθητών που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό δεν έχει μόνο ε, θετική επίπτωση ε, στην καταπολέμηση της πρόορης εγκατάλειψης σχολείου, αλλά σπάει και το φαύλο κύκλο που συνδέεται με τη φτώχεια και τις κακές επιδόσεις στο σχολείο. Περιμένω τις ερωτήσεις σας και τα επικοδομητικά σας σχόλια. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε τώρα στο γύρο με τη συζήτηση που θα ξεκινήσουμε. Ο κύριος Φίσα ζήτησε τον λόγο. Πρώτος παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και κυρίως θέλω να συγχαρώ τους τέσσερις εισηγητές για τις εισηγήσεις τους και κυρίως για την αξιόλογη δουλειά, πολύ αξιόλογη δουλειά που αναπτύσσουν. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι προς την ε, κυρία Χωτσικόβα, ότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ αξιοπερίεργη αυτή η τσεχική νομοθεσία αυτό αντί να προαχθεί η πρόθεση των ατόμων με ειδικές ανάγκες παρακολύεται η απασχόλησή τους μετά στις επιχειρήσεις. Στην Ισπανία έχουμε το αντίστροφο. Υπάρχει ένα νομοθέτημα, φοβούμαι δεν έχω τις λεπτομέρειες αυτού του νομοθετήματος, αλλά υπάρχει υποχρέωση των μεγάλων επιχειρήσεων και θεσμικών οργάνων να έχουν συγκεκριμένο αριθμό, ποσοστό των εργαζομένων τους με ειδικές ανάγκες και είτε είναι ε, διανοητική είτε σωματική αυτή η αναπηρία. Είναι υποχρέωση που έχουν ε, τα μεγάλα θεσμικά όργανα και οι μεγάλες επιχειρήσεις νομοθετικά στην Ισπανία και στην έδρα του κόμματός μας ε, του ε, Λαϊκού Κόμματος στη Μαδρίτη έχουμε ένα ε, παιδί, ένα νέο που ε, έχει μειονεξία και που στην υποδοχή των όσων προσέρχονται στα γραφεία του κόμματος αναλαμβάνει την διεκπαιρέωση αυτών των εργασιών και είναι ένας πολύ αγαπητός νέος σε όλους μας και σε σχέση με τις συναλλαγές με άτομα με ειδικέ ανάγκες και τις επαφές θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό να γίνεται αυτό και θα πρέπει να υποστηριχθεί αυτό σε σχέση με την ψήφιση για αυτά τα θέματα που ελπίζουμε ότι θα διευθετηθεί σύντομα. Για τα θέματα με ατόμων με ειδικέ ανάγκες και τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν και οι μετανάστες ε, και άτομα με ειδικές ανάγκες, ο αθλητισμός νομίζω προσφέρει δυνατότητες. Οι δυνατότητες που προσφέρονται από τον αθλητισμό είναι κάτι που έχει ε, δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί σε πολλές χώρες και είναι νομίζω σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Η κυρία Τρούπερ τώρα παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ Ντόρις. Θα ήθελα, αν γίνεται, να στραφώ στους εκπροσώπους ε, εισηγητές ή ότι και να πω ότι πολύ γοργά μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα διέξοδο με τις ε, ε, αρνητικές διακριτικές μετα... Ε, αντιμετωπίσεις των ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Το γνωρίζουμε αυτό ότι συμβαίνει. Αν μπορείτε να πείτε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα πώς καταφέρνετε εσείς να προσεγγίσετε νέους με διαφορετικές μειονεξίες και προβλήματα. Διότι όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα για νέους που δεν είναι πρόθυμοι να πηγαίνουν στο σχολείο, πώς μπορείτε να τους προσεγγίσετε, πώς μπορεί να δοθούν κίνητρα σε αυτά τα άτομα, πώς μπορεί να διασφαλιστεί μια κάποια συνέχεια να τονωθεί η αυτοπεποίθηση, ο αυτοσεβασμός, η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Ενδιαφερόμαστε να υπάρχουν τέτοια καλά παραδείγματα ως πρότυπα για να μάθουν οι άλλοι και να ακολουθήσουν αυτά τα πρότυπα. Θα ήθελα να ξέρω πώς δημιουργείτε τέτοιες επαφές και πώς μπορείτε να δώσετε κίνητρα σε τέτοιους νέους. Θα ήθελα να μου το απαντήσετε αυτό στην καθημερινή ζωή τι κάνετε. Ευχαριστώ. Uh, ναι. ah. Εγώ έχω τώρα σειρά. Και εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτά τα θέματα. Προσθέτω και εγώ την φωνή μου στα όσα είπε η Χέλγα Τρούπερ, η συνάδελφος πιο πριν. Πολύ σημαντικό θα ήταν αν είχαμε κάποια παραδείγματα παραπάνω. Το παράδειγμα από την Τσεχία είναι εξαιρετικό βέβαια και το weekend από την Ολλανδία ως παράδειγμα και αυτό πολύ καλό. Θα ήθελα να ξέρω πώς καταφέρνετε να πηγαίνουν οι νέοι στα ε, weekend groups αυτά. Τι κίνητρα δίνετε. Εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να εκπαιδευτούν προσέρχονται. Εκείνοι που δεν, ξέρουν τι θα κάνουν με τον ελεύθερο χρόνο τους έρχονται και αυτοί Πώς προσέρχεστε σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς τους προσεγγίζετε και τι κάνετε. Διότι έχει ένα επιπρόσθετο χαρακτήρα αυτό για εκείνους που ούτως ή άλλως ε, ε, βρίσκονται στην εκπαίδευση. Αναφέρθηκε ότι ε, θα ερχόταν και η κυρία Σάκερ. Καλό θα ήταν να παρίστατα να συζητούσαμε την πρότασή της, αλλά με άλλη εκδήλωση ή αφορμή θα συναντηθούμε και θα συζητήσουμε την πρότασή της. Για τον συνάδελφο, για τον κύριο Μαχίδη θα ήθελα να πω κάτι στο νεαρό κύριο Μαχίδη για τις προτάσεις σας για την αναγνώριση της μη επίσημης ε, εκπαίδευσης είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλές φορές εδώ και εδώ και πολύ χρονικό διάστημα. Σίγουρα στο μέλλον αυτό το θέμα των αλλαγών και των βελτιώσεων και της ε, προσοντοποίησης με το ευρωδιαβατήριο Europass ε, θα μας απασχολήσει ούτως ή άλλως. Είναι υπερβολικά αυστηρά ή περιορισμένο το φάσμα του στην επισημοποιημένη αν θέλετε παιδεία και εκπαίδευση. Και θέλουμε σε σχέση με τους νέους αυτό να είναι διάκριτο Αν θέλουν ε, και προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είναι πράγματα που και στην ε, Επιτροπή ε, την χάνουν σκέψεων και προβληματισμού και ο κύριος Σάνταν Ποκόνη είμαι βέβαια, ότι στα όσα θα μας πει θα μπορέσει να αναφερθεί σε αυτό το θέμα και για το Europass. Αυτά ήθελα να πω. Και τώρα η κυρία Χανίμπαλ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τους ε, ομιλητές μας που έκαναν πολύ ενδιαφέρουσες ε, εισηγήσεις. Εγώ θέλω να τονίσω αυτό που είπατε και εσείς, Πρόεδρε, και η κυρία Τρούπελ, ότι δυστυχώς όλα αυτά τελικά αφορούν το θέμα των πόρων. Όπως τα ξέρετε, είμαι ε, εισηγήτρια για την ε, έκθεση για την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου που μόλις την ολοκλήρωσα γιατί δυστυχώς δεν θα μπορέσω σε αυτό το στάδιο να ενσωματώσω τα όσα ακούσαμε τώρα αν και μπορεί και να τα προσθέσουμε με κάποιες τροπολογίες. Θέλω να σας ρωτήσω, όχι μόνο τι πόρους έχετε για σας και για τη δική σας δουλειά, αλλά και τι επιπλέον πόροι υπάρχουν για τους νέους με τους οποίους δουλεύετε. Ένας από τους λόγους για τους οποίους φεύγουν νωρίς από το σχολείο οι νέοι είναι οικονομικός. Αν δεν είναι πλούσιοι, ε, κοστίζει πολύ το να μείνουν στο σχολείο. Ξέρετε να υπάρχουν προγράμματα για οικονομική βοήθεια για τους νέους που θέλουν να μείνουν στο σχολείο. Και τι είδους πόρους έχετε εσείς για τη δουλειά σας. Συμφωνώ με την Πρόεδρο. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα παραδείγματα για το τι κάνετε. Αλλά με εντυπωσιάζει πάντα ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και εσείς οι ίδιοι κάνετε καταπληκτικό έργο. Αναρωτιέται κανείς τι γίνεται Ποιος κόσμος μπορεί να τα κάνει αυτά και αν υπάρχουν και αρκετά χρήματα για όλα αυτά. Και ίσως θα πρέπει να δουλέψουμε για ένα ευρύτερο σύστημα με καθολικές προβλέψεις για τον τομέα αυτό και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα ότι είναι λίγο μπαλώματα όλα αυτά που κάνουμε Τι οικονομική στήριξη υπάρχει λοιπόν για εσά και για τους νέους με τους οποίους δουλεύετε Θα επανέλθουμε στην κυρία Γκρίφιν, ήθελα να πω το εξής. Είπατε ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι κυρίως σε επαγγελματικά σχολεία. Και χαίρομαι γιατί έχουν εκεί τη δυνατότητα να βρουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους και να τις αναπτύξουν. Εξαρτάται βέβαια το πόσο καλή είναι αυτή η η επαγγελματική και πόσο οι ε, καθηγητές είναι προετοιμασμένοι. Εγώ δεν το καταγγέλω. Εσείς δεν ξέρω αν το καταγγείλατε ε, αυτό. Ίσως αυτό που φταίει και πρέπει να στιγματίσουμε είναι η εκπαίδευση των ε, καθηγητών. Χθε είπαμε και ο κύριος Μπίσκι και άλλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία οι νέοι μαθητές. Δηλαδή εκτός από την ανώτερη, ε, ανώτατη εκπαίδευση να μπορεί να πηγαίνουν και σε επαγγελματικές σχολές, να μαθαίνουν μια τέχνη, ένα επάγγελμα ε, που θα τους αποφέρει περισσότερα παρά να συνεχίσουν σε κάποιες άλλες ε, πνευματικά ανώτερες ατραπούς. Αυτό λοιπόν ε, που χωλαίνει νομίζω είναι η εκπαίδευση των δασκάλων και των καθηγητών. Και τι είναι η κυρία Χάνιμπαλ ότι είναι τόσο ακριβό το σχολείο. Δωρεάν θα πρέπει να είναι το σχολείο. Και η αξίωση να πηγαίνει κάνει σχολείο είναι δωρεάν. Δεν ξέρω, είναι ιδιαίτερα βρετανικό το παράδειγμα αυτό. Τι εννοείται ότι δεν έχουν χρήματα. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε κύριε Χάνιμπο. Ζητώ συγγνώμη. Ε, ίσως δεν το είπα καλά. Δεν είπα ότι κοστίζουν τα σχολεία. Οι επιπλέον εξωτερικές παρεμβάσεις και για τους μαθητές που φεύγουν από το σχολείο κοστίζει περισσότερο να παραμένουν στο σχολείο. Και πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο γιατί δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Έχουν ειδικά έργα, ειδικά project ε, οι καλεσμένοι μας σε αυτή την κατεύθυνση και παίρνουν και χρηματοδότηση. Η κυρία Μπέναραμπ, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. είμαστε στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του αποκλεισμού. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Χωράει μεγάλη ερμηνεία και πολλά πράγματα εντάσσονται. Και πριν έχουμε μια λίστα, ένα κατάλογο προγραμμάτων, πρέπει να έχουμε ένα πολιτικό όραμα. Και τι έχει σημασία για μένα, να προχωρήσουμε προς συστήματα που Ε, να έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, όχι να φτιάχνουμε πρώτα το σύστημα ε, για την πλειοψηφία και μετά ή την πλειονότητα και μετά η μειονότητα να καλείται να ενταχθεί. Γιατί ε, κινδυνεύουμε να έχουμε αποκλεισμούς γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των νέων και ψυχολογικές και εγώ είμαι από ένα φτωχό κοινωνικό στρώμα. Ο πατέρας μου ε, είναι εργάτης. Δεν είμαι γαλλόφωνη, η μητρική μου γλώσσα δεν είναι τα γαλλικά. Όταν ήρθαμε στη δεκαετία του 80 κατασταθήκαμε στη Λιόν, όπου υπήρχε μια κοινωνική ε, ε, πολυφωνία από ε, ε, διάφορες κοινωνικές προελεύσεις και φιλετικές προελεύσεις και ε, χώρες. Και, δηλαδή αυτό που μας χαρακτήριζε δεν ήταν η προέλευση κοινωνική, εργατική και μπορούσαν τα παιδιά να είναι κάτι άλλο από τους γονείς τους. τώρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και στην κοινωνία. Και είναι πάρα πολύ δραματικό. Θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικά συστήματα και το σχολείο βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή και το σχολείο θα πρέπει να αλλάξει πολιτική, όχι ο μαθητής να προσαρμοστεί στο σχολείο. Και στα διάφορα επίπεδα και στα κοινωνικά και στα σχολεία να είναι το σύστημα τέτοιο ώστε να επιτρέπει στον καθένα, ανεξάρτητα από την προέλευσή του ή από την ηλικία του ενήλικας ή παιδί, να εντάσσεται. Σήμερα υπάρχουν οι νέες τεχνολογίες που το επιτρέπουν για παράδειγμα, με τους υπολογιστές μπορούν οι τυφλοί να έχουν πρόσβαση ε, σε υπολογιστές. Να, να γίνεται με όραμα όμως. Να ανοιχτά τα συστήματα, ε, να σέβονται τη διαφορετικότητα του καθενός και όχι να έχουμε ένα σύστημα κορσέ όπου θα πρέπει ο καθένας να φροντίσει να χωρέσει εκεί μέσα. Αυτά. Να μην είναι το σχολείο ένα καλούπι, πούμε. Σε σχέση με το όσο είπε η κυρία Μπροζίκοβα από τη Τσεχία. Είπε ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν συνεισφέρουν ποτέ στην ευημερία μιας χώρας. Μα για μένα αυτό είναι εξωφρενικό. Φυσικά και μπορεί ο καθένας να συνεισφέρει στην ευημερία. Τι θα πει ότι είσαι απροσάρμοστος απροσάρμοστο με βάση το σύστημα που σου επιβάλλει να μπει στο καλούπι αυτό. Όχι, θα πρέπει να είναι ανοιχτό και να προσαρμόζεται το σύστημα στον κόσμο. Ευχαριστώ. Κυρία Μπεναράμπ Ατού. Απαντήσεις. Η κυρία Μπροζίκοβα πρώτη. Όχι, με την αντίστροφη σειρά τώρα οι απαντήσεις. Ο κύριος Μαχίδη πρώτος και μετά οι υπόλοιποι. Μουράτ Μαχίδη. Ευχαριστώ αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα αναφέρθηκαν. Θα προσπαθήσω να ταξινομήσω τη σκέψη μου σε σχέση με αυτέ τις παρατηρήσεις. Αυτό που ρώτησε η κυρία Τρίπελ, πώς μπορεί να τονωθεί η αυτοπεποίθηση, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα άτομα με μειονεξίες από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Είναι λοιπόν σημαντικό σε σχέση με τις ε, οργανώσεις νέων. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα αυτό, διότι πολύ συχνά βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να πάμε προς αυτούς, ε, να κινηθούμε προς αυτούς. Αυτό όμως που διαπιστώνουμε είναι ότι αυτή η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, η συμμετοχή αυτή είναι κάτι που το μαθαίνει κανείς από την παιδική ηλικία και όσο νωρίτερα ξεκινάμε σε ηλικιακά, σε ε, πρώιμη παιδική ηλικία, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία αυτούς τους νέους στο τέλος να τους εντάξουμε στις οργανώσεις νέων και να τους προωθήσουμε ώστε να ενταχθούν κοινωνικά και εργασιακά. Ωστόσο όμως πάντα δεν είναι τόσο εύκολο να γίνεται αυτό. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας πολλές φορές μεταξύ των οργανώσεων νέων και των κοινωνικά μειονεκτικών ομάδων. Και αυτό ξεκινά ήδη από τις οικογένειες και πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα σε σχέση με το να μπορέσουμε να πετύχουμε την ένταξη αυτών των νέων. Ένα πρόβλημα που πολύ συχνά βλέπουμε να υφίσταται είναι πόσο συχνά στο τέλος οι οικονομικές ε, προϋποθέσεις και συνθήκες διαδραματίζουν ένα ρόλο που χρειάζεται μεγάλη υποστήριξη για την ένταξη αυτών των νέων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το χάσμα, να γεφυροποιήσουμε αυτό το χάσμα, να κάνουμε δουλειά με τους νέους, να συναντούμε τους νέους και τα παιδιά εκεί που ζουν και βρίσκονται και ε, ε, έχουν γεννηθεί και όχι να περιμένουμε να προσέλθουν αυτά τα παιδιά και να νέοι σε εμάς οι ίδιοι, να πάμε εμείς σε αυτούς και αυτό το οποίο αναφέρθηκε σχολεία επαγγελματική κατάρτισης. Έχετε δίκιο ότι αυτό δεν είναι καταρτικό. Αυτό το οποίο όμω είναι σημαντικό για μα είναι ότι δεν πρέπει να είναι προκαθορισμένο κοινωνικά ποιο παιδί θα πηγαίνει σε ένα τέτοιο σχολείο επαγγελματική κατάρτισης και ποιο θα πηγαίνει στην ανώτερη εκπαίδευση, βαθμίδα εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα κάνει να δίνουμε ευκαιρίε στους νέου να επιλέξουν οι ίδιοι, να επιλέξουν οι ίδιοι οι νέοι ποια σταδιοδρομία, ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν δεν επιτρέπεται, δεν είναι δυνατόν τα φτωχά ε, παιδιά να καταλήγουν στα σχολεία επαγγελματική κατάρτιση και τα άλλα πιο πλούσια, πιο ε, παιδιά από πιο ευκατάστατε οικογένειε να μπορούν να συνεχίσουν ε, σε, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιε έντονε, τέτοιε μεγάλε ανισότητε. Και μια άλλη σκέψη που θέλω να σα εκθέσω Εκείνο το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ τη συμμετοχή και ένταξη των παιδιών είναι η γκαιτοποίηση. Όταν οι κοινωνικέ ομάδε δεν έχουν επαφή μία με την άλλη και βρίσκονται στεγανοποιημένε, περιθωριοποιημένε η μία δίπλα στην άλλη, τότε δυσχεραίνονται πολύ τα πράγματα. Και σε σχέση και μία ε, οργάνωση νέων που ε, αν δεν βρισκόταν στην περιφέρεια στην, ε, στην οποία ζούσα ή στη συνοικία στην οποία ζει κάποιος για παράδειγμα αυτό δημιουργεί προβλήματα και έτσι αυτό, η οικετοποίηση αυτή η στεγανοποίηση δημιουργεί πρόσθετο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα θέλαμε να ξέρουμε τώρα πώς τα καταφέρνετε εσείς, πού ξεκινάτε και πώς το κάνετε. Η εγκαιτοποιηση αυτη η την περιγραφή του προβλήματος τη γνωρίζουμε και πως το κανετε η περιγραφη την περιφερεια του προβληματος τη γνωριζουμε και μπορουμε να την κάνουμε και εμείς. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε ξέρουμε συγκεκριμένα χειροπιαστά τι κάνετε εσείς στην οργάνωσή σας. Πώς βρίσκετε αυτούς τους νέους και πώς τους προσεγγίζετε και τι κάνετε. Για την περιγραφή μπορεί κανείς να το κάνει οποιοδήποτε. Αλλά τέλος πάντων δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Η κυρία Τερβέν παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω συγκεκριμένα να απαντήσω. Πώς φτάνετε στους νέους. Από την ηλικία των 10 ετών και μάλιστα σπρώχνονται για να έρχονται στο σχολείο του Σαββατοκύριακο. Ε, πώς γίνεται αυτό, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Μια στιγμή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σύμφωνα με τις έρευνες, ε, οι νέοι που εγκαταλείπουν το σχολείο, drop out, λένε ότι δεν θέλω να πάω ε, στο σχολείο γιατί δεν με αφορά το σχολείο. Δεν ξέρω τι θα μου αποφέρει, δεν με ενδιαφέρει και τι θα έχω από αυτό. Αυτό είναι χρήσιμο και ωραίο να το έχουμε στο μυαλό μας για τέτοια προγράμματα όπως είναι το σχολείο του Σαββατοκύριακου γιατί το θέλουν οι νέοι. Τους αρέσει. Όταν πας και τους λες κοίτα έχουμε αυτή την προσφορά, σε ενδιαφέρει, τους ενδιαφέρει και έρχονται. Σηκώνουν το χέρι τους όλοι και γράφονται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουμε νέους, το πρόβλημα είναι ότι έχουμε λίστες αναμονής και δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε. Θέλουν όλοι να έρθουν στο σχολείο μας. Αυτό ως πρώτο σημείο, ε, γιατί οι νέοι θέλουν να μαθαίνουν τα παιδιά, οι μαθητές ενδιαφέρονται να μαθαίνουν, αλλά να μαθαίνουν κάπου που τους ενδιαφέρει και να θεωρούν ότι τους αφορά αυτό που μαθαίνουν. Συμφωνώ πολύ με το γείτονά μου ε, το παρακαθήμενο ότι οι οργανώσεις νέων, η συλλογικότητα είναι κάτι το οποίο μαθαίνει στα παιδιά πάρα πολλά πράγματα αλλά ακριβώς ε, στην ηλικία των 10 ετών είναι πολύ νωρίς. Βεβαίως η εμπειρία του σχολείου μας ε, ε, αποδεικνύει ότι τονώνει την αυτοπεποίθησή τους. Κάθε Κυριακή έρχονται, ε, δηλώνουν θελοντικά για τα επόμενα προγράμματα και τα ενδιαφέροντα που τους προσφέρουν. Και έχουν και προθυμία και όρευση, θέλουν να συμμετέχουν. Η ηλικία 10 ετών δεν είναι τυχαία, είναι προεφηβική, είναι καλή στιγμή να τους κάνεις να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα και θέματα που τους ενδιαφέρουν και πραγματικά αποδίδει. Κάποιος μίλησε για την άτυπη εκπαίδευση, την ανεπίσημη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για την πολιτική. Βέβαια, εγώ πολιτικός δεν είμαι, αυτό είναι δική σα δουλειά, αλλά θα πρέπει να ε, διατηρηθεί η διάκριση ε, της εκπαίδευσης της επίσημης κλασικής, τι πρέπει να μάθει στους νέους, ε, να διαβάζουν, να γράφουν, να υπολογίζουν μαθηματικά, ωραία όλα αυτά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά και δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο. Πέρα από την επίσημη λοιπόν εκπαίδευση θα πρέπει να μάθουν και πάρα πολλά πράγματα. Και ποιο είναι το ωραίο εδώ. Αυτή η άτυπη εκπαίδευση είναι κάτι που ενδιαφέρει και την κοινωνία και εδώ ενδιαφέρον αυτό από πλευρά οικονομικού κόστους και οι επιχειρήσεις ας πούμε προτείνουν ε, περιόδους άσκησης, μαθητεία, στάζ για τους νέους ε, σε όλους τους ε, τομείς. Και η πολιτική επιλογή εδώ θα είναι να υποστηριχθεί αυτό για να γίνεται. Εμείς στην Ολλανδία τι βλέπουμε. Ότι η επίσημη εκπαίδευση, το επίσημο σχολείο αποτυχάνει πολλές φορές. Δηλαδή μαθητές παρόλο που πηγαίνουν στο σχολείο δεν ξέρουν ούτε να διαβάζουν, ούτε να γράφουν, ούτε να ε, λογαριάζουν. Και ακριβώς στις άτυπες μορφέ εκπαίδευση ενδιαφέρονται και συμμετέχουν πάρα πολύ. και είμαι πεπισμένη εγώ από την εμπειρία μου. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν μας θέλουν οι μαθητές, ότι εμείς ε, θα πρέπει να τους προσελκύσουμε, να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες οι δικές μας προτάσεις και προσφορές. Και ποιος θα πληρώνει όλα αυτά. Μα ακριβώς εκείνη το κλειδί, η κοινωνία των πολιτών. Και ε, τα χρήματα που διοχετεύονται στη δημόσια εκπαίδευση να πηγαίνουν ακριβώς προς την κατεύθυνση που χρειάζονται οι νέοι. Εμείς πώς χρηματοδοτούμε τη δουλειά μας, το είπα προηγουμένως, ε, από ιδιωτικές επιχειρήσεις, εταιρείε που ενδιαφέρονται πάρα πολύ ε, σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρίφιν τώρα. Um, and thank you for the... Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τα σχόλια που νομίζω ε, ήταν πολύ κέρια. Μας ρωτήσατε αν υπάρχουν πρακτικές, ε, πρακτικά παραδείγματα για τα όσα συμβαίνουν. Σας αναφέρω τα εξής. Το, το θέμα για το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα, το κόστος του να μείνει κανείς στο σχολείο είναι κάτι το οποίο έχει αναγνωριστεί. Ιδιαίτερα για τους πολύ καλούς μαθητές που κανείς μπορεί και να ελπίζει να πάνε και στο τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εγώ ασχολούμαι με το πρόγραμμα ε, του Δυτικού Δουβλίνου σε μια ιδιαίτερα μεικτονεκτούσα περιοχή. Συνεργαζόμαστε με τους φοιτητές εκεί, τους μαθητές εκεί και να μπορέσουμε να τους διευκολύνουμε να φτάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό που λειτουργεί καλά, από ό,τι έχουμε δει από την εμπειρία μας, είναι η πρόσβαση σε κάποια υποτροφία. Αν μείνουν δηλαδή και μετά το σχολείο και μελετούν και φοιτούν για ένα χι αριθμό ε, μαθημάτων παραπάνω μέσα στην εβδομάδα, παίρνουν μία υποτροφία. Δεν είναι πολλά χρήματα, αλλά ε, τους ε, τραβάει. 15 χρόνια δουλεύει τώρα αυτό το σύστημα και η ε, βέβαια, μειώνεται διαρκώ η υποτροφία γιατί η παράδοση πρόσβαση στο ειδοβάθμιο εκπαίδευση έχει πλέον ε, ε, εμπεδοθεί μέσα στην κοινότητα. Αυτό το σύστημα λοιπόν λειτουργήσε πολύ καλά. Κάποιο άλλο ανέφερε την κατάρτιση των εκπαιδευτών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί περισσότεροι δάσκαλοι όταν πηγαίνουν σε κάποια κολέγια κατάρτιση ε, μαθαίνουν πώς να διδάσκουν ακαδημαϊκά θέματα, αλλά δεν μαθαίνουν ε, γενικά να διδάσκουν στα άτομα με ειδικέ ανάγκες που είναι στις τάξεις τους, ούτε για να χειριστούν τα παιδιά μεταναστών με τεράστιες ροές που πολλές φορές δεν ξέρουν καν να μιλάνε τη γλώσσα του σχολείου δεν μαθαίνουν ε, πώς να αντιμετωπίσουν τους, ε, τα παιδιά που έχουν κοινωνικά προβλήματα ε, το θέμα λοιπόν της διαρκούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτών είναι πολύ σημαντικό Χρειάζεται ειδική κατάρτιση για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και ε, ειδική κατάρτιση για την διδασκαλία της γλώσσας, να είναι πιο αποτελεσματικές οι διδασκαλίες. Δηλαδή, δεν είναι ότι ο κόσμος πρέπει να κατηγοριοποιηθεί. Έχουν δικαίωμα όλοι σε ποιοτική εκπαίδευση. Οπότε, η κατάρτιση των εκπαιδευτών είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλοι, λοιπόν, όταν θυμούνται το σχολείο τους, θυμούνται ποιοι οι δάσκαλοι τους επηρέασαν και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τα παιδιά από τις μειονεκτούσες περιοχές. Γιατί ένας από τους λόγους που αφήνουν το σχολείο είναι γιατί λένε ο δάσκαλος δεν με ήθελε, δεν με συμπαθούσε. Η αυτοπεποίθησή τους είναι τόσο χαμηλή που αν κάνει ένα λάθος σχόλιο ο δάσκαλος μπορεί το παιδί να παρατήσει το σχολείο. Η δουλειά λοιπόν με τους ίδιους τους εκδιδάσκαλους είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το συναισθηματική πτυχή της διδασκαλίας που είναι πάρα πολύ σημαντική και ακόμη πιο σημαντική για τα παιδιά από σε περιοχές. Τώρα όσον αφορά την άτυπη, την ανεπίσημη παιδεία έχουμε διάφορα προγράμματα ιδιαίτερα για τα παιδιά πάνω των 16 ετών και έχουμε ένα πάρα πολύ αποτελεσματικό για τα παιδιά κάτω των 16. Δηλαδή στο μετέχμιο. Ο συνάδελφος έχει δίκιο. Πρέπει να γίνουν πιο πρακτικά θέματα μαζί τους για να ασχοληθούν. Δηλαδή η δουλειά η ξυλουργού, Ε, ο συνάδελφος από την Ισπανία είπε, είπε ότι ο αθλητισμός πολύ συχνά τραβάει τα παιδιά οποιοδήποτε δεσμό μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να κρατήσεις τα παιδιά στο πρόγραμμα. Το δύσκολο είναι ότι έχουμε τόσο λίγα χρήματα για τέτοιου είδους προγράμματα που και πάντα πρέπει κανείς να εξισορροπήσει τα πράγματα για να δει πού θα πάει. Δηλαδή είναι λίγο... Είναι δύσκολο να, να αποφασίσεις ποιος θα πάρει τι. Γιατί σε σχέση με τη βασική και κανονική εκπαίδευση τα επιπλέον χρήματα είναι ελάχιστα. Αλλά ακόμα και ένα ελάχιστο ποσό μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο. Γιατί όταν μιλάμε για τα παιδιά τους, φοιτητές, τους μαθητές ε, που χρειάζονται περισσότερο, τους, τα, τους μαθητές που προσπαθούμε να τους κρατήσουμε έξω από τις αντικοινωνικές δραστηριότητες, δηλαδή στην ουσία προσπαθούμε να τους κρατήσουμε έξω από τις φυλακές, είναι μικρός αριθμός παιδιών και λίγα χρήματα μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν προγράμματα λοιπόν που λειτουργούν αποτελεσματικά και που θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα αν είχαν περισσότερα χρήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και τέλος η κυρία Μπροσίκοβα. Θα ήθελα καταρχάς να απαντήσω ε, στα όσα είπε η κυρία Ευρωβουλευτής από τη Γαλλία ε, για ε, τα άτομα με μέτρια ή σοβαρή διανοητική αναπηρία και κατά πόσο μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας ή στην ηθική εξύψωση μπορούν να συμμετέχουν. Βεβαίω, σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο Ισπανός Ευρωβουλευτής, οι ε, εργοδότες έχουν την υποχρέωση να ε, προσλαμβάνουν ε, άτομα με σωματική αναπηρία ε, που να μπορούν όμως να εργαστούν. Αυτό δεν ισχύει πάντα ε, ε, με εκείνους που πάσχουν από το σύνδρομο down. Ούτε μπορεί ο κάθε εργοδότης να προσλαμβάνει τέτοια πρόσωπα ούτε είναι διατεθειμένος να ε, πληρώνει ε, υψηλούς φόρους σε εισφορές ή να έχει ε, ειδικέ θέσεις απασχόλησης προστατευμένες και αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία που έχουν διάφορα εργαστήρια και παράγουν διάφορα προϊόντα. Πολλές φορές επιλέγουν τις εύκολες λύσεις οι εργοδότες. Υπάρχει μια τάση επίσης να παραμένουν να κρατούνται οι μαθητές στο σχολείο μέχρι την ηλικία των 15 ή 17 ετών, ακόμα και αν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, να μένουν στην ίδια τάξη. Ή τα παιδιά των μεταναστών που φοιτούν στα σχολεία, τα εγκαταλείπουν πρόωρα. Υπάρχουν επίσης προβλήματα με τους Ρωμά ε, που λατρεύουν την ελευθερία τους και δεν, θέλουν δεν τους αρέσει να πηγαίνουν σχολείο. Αν όμως κανείς δεν... Αν δεν πηγαίνουν μάλλον τα παιδιά αυτά σχολείο, αφαιρούν από τους γονείς τους ε, ε, τα οικογενειακά επιδόματα και τα επιδόματα τέκνων οι αρχές. Οπότε παραμένουν τα παιδιά στο σχολείο μέχρι την ηλικία των 15 και των 17 ετών. Ευχαριστώ. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Μιλήσατε για ένα νέο που ήταν τόσο καλός και τόσο επιμελής και τόσο τα κατάφερνε και δεν έβρισκε δουλειά. Μα αν υπάρχει αυτός ο νόμος, όπως είπε ο κύριος Φίσας, γιατί δεν τον προσλαμβάνουν τα εργοστάσια, οι εργοδότες, διότι ο τσεχικός νόμος απαιτεί να είναι ο ε, εργαζόμενος σε θέση να βάλει την υπογραφή του. Ε, ε, α, είναι αντίφαση αυτό λέει η κυρία Πάκνα, γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασία του σχολείου με την επιχείρηση για να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση για τους μαθητές αυτούς που πάσχουν από σύνδρομο Down για να εργάζονται ε, σε διάφορες επιχειρήσεις κάποιων επιχειρηματικών κλάδων. Εμείς ζητήσαμε να αλλάξει η νομοθεσία. Σας είπα ότι είχαμε την εμπειρία με τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στην Ιταλία, ε, όπου οι μαθητές, οι σπουδαστές μπορούν να εργάζονται ε, χωρίς να είναι υπεύθυνοι διανόμου και να υπογράφουν ε, τη σύμβασή τους με την επιχείρηση. Και ακόμα ε, και αν δεν έχουν περάσει τις συναγωγικές εξετάσεις και δεν έχουν επιτύχει. Αυτό είναι διαφορά στην νομοθεσία. Ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή ευρωπαϊκή νομοθεσία για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κυρία Τρούπερ, θα ήθελε να αναφέρει κάτι για ένα παραδείγμα και ο κύριος Ποκόρνη μετά θα λέει τον λόγο. Θα ήθελα να δραχθώ τη ευκαιρία να σας αναφέρω δύο, όπως πιστεύω, πολύ πιστικά παραδείγματα πώς ε, το έργο της εκπαίδευσης παιδείας ε, με τους νέους ε, και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να στεφθεί με επιτυχία. Από τη δική μου περιοχή στην Βρέμη, στην Ομοσπονδική Γερμανία. Υπάρχει μια ορχήστρα, η Φιλαρμονική της Βρέμης, που ανήκει στις 10 καλύτερες ορχήστρες του κόσμου παγκόσμια και που μετακόμισε σε ένα κοινωνικά μειονεκτικό, σε μια μειονεκτική συνοικία και εργάζεται με τους νέους, δίνει τα όργανα για να μπορέσουν να, ε, παίξουν οι νέοι και διοργανώνει συναντήσεις ώστε στη συνοικία αυτή άλλοι ε, οικοί και φίλοι και συγγενείς να μπορέσουν να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν αυτές τις συναυλίες. Έχουν κάνει εξαιρετικέ ε, εμπειρίες, διότι ενισχύει, τονώνει την αυτοπεποίθηση των νέων, η δυνατότητα αυτή ε, να ενασχοληθούν με τη μουσική, κάτι που δεν είχαν προηγούμενα ως δυνατότητα. Ένα παράδειγμα που δείχνει πώς η εγκατάσταση ενός σχολείου με τη δραστηριότητα μιας ορχήστρας σε μια συνοικία δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης των μειονεξιών και σε σχέση με μια ε, ορχήστρα που δεν επιλέγει την πιο πλούσια συνοικία για να δραστηριοποιηθεί αλλά δρά με αυτόν τον τρόπο. Το άλλο πρόγραμμα ονομάζεται Blaumeier. Ξεκίνησε από ένα ψυχιατρικό πρόγραμμα. Δουλεύει εδώ και 25 χρόνια με άτομα με το σύνδρομο Down, με σχιζοφρένειες, με κατάθλιψη, μανιοκατάθλιψη, με ε, σωματικές μειονεξίες και άλλες. Έχουν ατελεία σεμινάρια τέχνης, έχουν παράξει ήδη ταινίε που έχουν γυρίσει και βρέθηκε απήχηση σε όλη την πόλη όπου άτομα με μειονεξίες και άτομα χωρίς μειονεξίες συνεργάζονται. Για παράδειγμα σε αυτή την ε, ε, έκθεση τέχνης, ε, σε μια αίθουσα τέχνης εκθέτουν πίνακες, καλλιτεχνική δουλειά τους, οικαστικά που έχουν με αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουν ενώ προηγούμενα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Δεν ήθελα να προσθέσω λέει Πρόεδρος και εγώ το εξή. Αυτό που πρέπει να πετύχουμε με όλους τους νέους είναι αυτά τα τέσσερα πράγματα. Το να να γνωρίζουν κάτι, να γνωρίζουν να κάνουν κάτι, να γνωρίζουν να είναι κάτι και να γνωρίζουν να μάθουν να συμβιώνουν. Αυτά είναι τα τέσσερα σημαντικότερα πράγματα που σε όλα τα επίπεδα πρέπει να πετύχουμε και να καταφέρουμε. Είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα, αλλά αξίζει τον κόπο. Και τώρα ο κύριος Άνταμ Ποκόρνη θα λάβει τον λόγο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μετά από αυτή την εισαγωγή, εγώ πώς να σταθώ στο ύψος σας. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε κάποιου περιορισμού βεβαίω στο πεδίο δράση μα και ανάληψη πρωτοβουλειών. Αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, Μπορούμε να κάνουμε πολλά με χρηματοδότηση προγραμμάτων, ιδιαίτερα την νεολαία σε δράση, τα διαρθρωτικά ταμεία, τη διαβίου μάθηση και πολύ περισσότερο βοηθώντας τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται και από, να ε, διδάσκονται από βέλτιστες πρακτικές αμοιβαία σε πολλά από αυτά τα κρίσιμα θέματα. Ευχαριστώ όλους τους σήμερα. Μας έδωσαν πολύ ε, σημαντικές και χρήσιμες ε, προτάσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνεται η πολιτική σημασία. Αν κοιτάξτε τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και τη συγκρίνεται με τη στρατηγική της Λισαβόνας, μία από τις μεγάλες διαφορές είναι η κεντρική ιδέα και θέση που δίνεται τώρα σε θέματα ισοτήτων ευκαιριών στην εκπαίδευση και στη συμπερίληψη. Δύο από τους έξι στόχους για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για την εκπαίδευση και ο ένας είναι για τα ε, ε, συστήματα που να προωθούν τις ευκαιρίες και να μειώνουν την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου. Και ο λόγος γι' αυτό είναι πολύ, ε, βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικός και κοινωνικός. Οι κοινωνίες μας είναι ε, πολύ πολιτισμικές, ποικιλόμορφες, ε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήνουμε ταλέντα και ικανότητες και δεξιότητες να πηγαίνουν χαμένα ε, λόγω κοινωνικής προέλευσης. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο στο οποίο εργαζόμαστε στην Ευρώπη, ε, τα θέματα που σας απασχολούν. Αν μου επιτρέπετε να επανέλθω σε ένα θέμα που έθεσε η κυρία Γκρίφιν όταν είπε ότι στην Ελλανδική νομοθεσία υπάρχει αυτό το κενό ως προς τα κονδύλια και τους πόρους που υπάρχουν. Βεβαίως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε σε εποχές οικονομικής κρίσης τόσο ακριβά συστήματα, αλλά το κόστος της μη αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος στην κοινωνία αργότερα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Όταν φεύγουν και εγκαταλείπουν το σχολείο πολλοί νέοι θα έχουμε πολύ μεγάλο κόστος και για τη δικαιοσύνη και για την υγεία και για την απασχόληση από ε, το εάν το προλαμβάναμε. Και αν θεωρεί κανείς ότι είναι ακριβή η ε, ε, παιδεία, ας δοκιμάσει πόσο ακριβή είναι η άγνοια η αμορφωσιά. Και μπορεί αυτό το θέμα να εμφανίζεται ως θέμα ε, παιδείας είναι πολύ ευρύτερο. Τα αίτια και ε, η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά ε, με εκπαιδευτικές μεθόδους ή με ε, λύσεις από πλευράς παιδείας. Θα πρέπει πολύ να μας απασχολήσουν ορισμένα από τα παραδείγματα που μας είπε η κυρία Τρίπελ. Με ποιο τρόπο θα κάνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν, όχι μέσω της κλασικής επίσημης ε, εκπαίδευσης. Θα ήθελα να αναφέρω μερικούς τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούμε. Το ένα ακούστηκε πολλέ φορέ είναι η πρόληψη τη ε, προώρης εγκατάλειψη σχολείου. Το Συμβούλιο Υπουργών την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε μια σύσταση που τόνισε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε συνεκτικέ συνολικέ στρατηγικέ που να καλύπτουν όχι μόνο την παιδεία αλλά και θέματα κοινωνικά, υγείας, ε, κοινωτική πολιτικής, ε, διαβίου μάθησης κτλ. Επίσης τονίζουμε τη σημασία της μέτρησης και της ανάλυσης κατάστασης σε πολλές χώρες. Είναι άγνωστη η κατάσταση πότε και γιατί φεύγουν νωρίτερα οι μαθητές από το σχολείο, πώς είναι αυτοί και σε περιφερειακό επίπεδο και επίσης ε, ποιες είναι εκείνες οι παρεμβάσεις που είναι ε, οι πιο αποτελεσματικές. Η αποτελεσματικότερη είναι η πρόληψη. Και αυτό έχει να κάνει με την αποφύγη κάποιων εξαναγκασμών να πηγαίνουν σε ένα σχολείο που δεν θέλουν ή που δεν τους ταιριάζει ε, οι μαθητές να υπάρχουν και άλλες μορφές σχολείων, όπως τα σχολεία για το Σαββατοκύριακο που ακούσαμε, πολύ σημαντικό, πολύ χρήσιμο, ο πολιτισμός, αθλητικές διοργανώσεις, ε, να ενθαρρύνονται ε, οι νέοι και οι μαθητές να μαθαίνουν από δραστηριότητες που δεν μοιάζουν εκπαιδευτικές εκ πρώτης όψεως. Και στην Ιρλανδία υπάρχουν καλά παραδείγματα. Με πολύ σημαντικό περιεχόμενο να καταλάβει κάποιος ότι είναι πολύτιμη η μάθηση και όχι κάτι που κάνει για ένα σχολείο ή για ένα καθηγητή επειδή στο ζητάει και είσαι υποχρεωμένο. Προσβλέπουμε στην έκθεση κυρία Χάνιμπολ της Επιτροπής σας και θα καλέσουμε σε μια ομάδα εργασία στα κράτη-μέλη να συνοδεύσουν την εφαρμογή αυτής της σύστασης. Δεύτερο σημείο. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που δεν αναφέρθηκε σήμερα, και αυτό είναι ε, παράδοξο, είναι η, προωρή, η νηπιακή ε, κατάρτιση και φροντίδα, γιατί όσο νωρίτερα μπουν τα παιδιά στην παιδεία, τόσο περισσότερο μένουν στο σχολείο και καλύπτουν τα μειονεκτήματα. Ε, Σαφώς η προηγούμενη έκθεση κύριε Χάνιμπολ που το αναφέρει αυτό και εγκρίθηκε πρόσφατα ε, το τονίζει. Δηλαδή πρέπει το σύστημα να είναι προσβάσιμο. Πώς δηλαδή φέρνει τον κόσμο, αλκύει τον κόσμο. Δηλαδή οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι άνθρωποι που το χρειάζονται περισσότερο να έχουν πρόσβαση, να είναι ελκυστικά τα σχολεία, τα ανεπινυπιακή σταθμή, ακόμα και σε αυτούς που δεν ε, αισθάνονται μεγάλη αυτοπεποίθηση για να μπουν στα επίσημα συστήματα. Η παρέμβαση αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ ψηλή ποιότητα, γιατί διαφορετικά μπορεί να είναι βλαβερή. Και αν όντω είναι ψηλή ποιότητα, ε, η απόδοσή τη είναι εντυπωσιακά ψηλή. Τρίτο τομέα είναι η ένταξη των μειονοτήτων και των μεταναστών. Και για τους Ρώμα, όπως ξέρετε, είχαμε ένα πράσινο βιβλίο το 2008 για το θέμα αυτό Τώρα ετοιμάζουμε ένα δίκτυο πολιτικής για, με χρήση του προγράμματος διαβίου μάθησης για να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τα συστήματα μας να γίνουν πιο ευέλικτα. Αυτή είναι μια πρόκληση που αναφέρθηκε για το πώς δηλαδή τα εκπαιδευτικά συστήματα μπορούν να απορροφήσουν την αυξημένη και αυξανόμενη διαφοροποίηση των μαθητών που έχουν. Ε, πώς τα σχολεία και οι δάσκαλοι και οι σχολικές δομές θα μπορέσουν να προσφέρουν ένα, σε, σε όλον τον κόσμο ε, την ευκαιρία να πετύχουν από όποιο περιβάλλον και προέρχονται οι μαθητές. Και αυτή είναι τεράστια πρόκληση για τους Ρώμα. 10 ε, εκατομμύρια είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ένωση και πιθανότατα η πιο μειονεκτική μειονότητα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα υιοθετήθηκε η στρατηγική για τους Ρωμά στην Κομισιόν με ένα μεγάλο κεφάλαιο για την παιδεία. Πρώτος στόχος είναι το να τελειώνουν το δημοτικό σχολείο. Πολλά παιδιά δεν τελειώνουν καν αυτό. Και βέβαια και η Ρώμα, όπως και για τους υπόλοιπους πληθυσμούς, θα πρέπει να στοχεύσουμε τις ανάγκες τους για να μπορέσουν να προσχωρήσουν και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Κομισιόν μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια εφαρμόζουν μια πρωτοβουλία για να καταρτήσουν χίλιους διαμεσολαβητές Ρωμά που θα κάνουν το σύνδεσμο ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και τι κοινότητε των Ρωμά για να μπορέσουν να ελκύσουν τα παιδιά των Ρωμά. Επίσης, θα γίνουν και ειδικά προγράμματα με μισό εκατομμύριο ευρώ είναι, προβλέπεται για αυτά για να εξερευνηθούν οι τρόποι προσέλκυσης των μαθητών στα σχολεία. Επίσης, ε, του χρόνου προβλέπουμε τα εξής. Ανακοίνωση για την παιδεία και την αναπηρία και την ένταξη. Αυτό θα εξετάσει τις, ε, την παιδεία για τα άτομα με δικές ανάγκες, ίσως ε, ε, την κατάρτιση των δασκάλων, πώς τα συστήματα μπορούν να απευθύνονται σε περισσότερο κόσμο και κάτι που αναφέρατε εσείς, Πρόεδρε, να εξετάσουμε το ευρύτερο πεδίο δεξιοτήτων που πολλές φορές ναι μαθαίνει κανείς στο σχολείο αλλά και εκτός σχολείου σε, άτυπη, σε άτυπο περιβάλλον και πώς ε, τα μέσα όπως το Europass και άλλοι ε, είναι πιο ευέλικτα και να αναγνωρίζουν καλύτερα τι έχει μάθει ο κόσμος, γιατί η παιδεία, η μάθηση καμιά φορά ε, και σε μεγάλο βαθμό πλέον αποκτάται εκτός των σχολικών συστημάτων. Και όσον αφορά τώρα τη χρηματοδότηση. Εμείς ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να εξετάσουμε μαζί με το Συμβούλιο και το, και το Κοινοβούλιο είναι πώς η χρηματοδότησή μας θα είναι πιο αποτελεσματική για το χειρισμό αυτών των θεμάτων. Λόγω τώρα των θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμο τρόπο αντιμετώπισης της μειονεξίας, ε, θα πρέπει να δούμε πέρα και από την παιδεία, δηλαδή να συνδυάσουμε και άλλους τομείς και το περιφερειακό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό και θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί εσείς εφήβρατε αυτή τη δράση, το ΡΕΤΖΙ, με, είχε υπέροχα αποτελέσματα τη διάσκεψη την περισμένη εβδομάδα μόλις έγινε για τα προγράμματα Regio, μια μεγάλη διάσκεψη. Ο, εκεί πολύ ουσιαστικά θέματα συζητήθηκαν για τα σχολεία, ε, για τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλους τομείς όπως η άθληση, ο αθλητισμός, κοινοτικές, ε, ε, κοινοτική εργασία, αστυνομική εργασία, η ανταπόκριση στην αντικοινωνική συμπεριφορά, η ένταξη, το πεδίο είναι τεράστιο και το δυναμικό είναι επίσης σπουδαίο και γι' αυτό και η περιφερειακή δράση πραγματικά βλέπουμε ότι ε, κάνει διαφορά. Και έπειτα, όσο νωρίτερα παρέμβει κανείς τόσο καλύτερο. Οι δεύτερε ευκαιρίε θα πρέπει να θεωρηθούν τελευταίο τελευταία λύση και κάτι στο οποίο στρέφονται τα σύστημα αν δεν έχουν καταφέρει να προλάβουν. Η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία και η σχολική ηλικία είναι το κλειδί και αυτό αναγνωρίζεται όλο ένα και περισσότερο σε επίπεδο της Ένωσης. Υπάρχουν προγράμματα όπως το Κομένιος και το μελλοντικό πρόγραμμα ε, για την παιδεία θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάνταμ. Πολύ ωραία όλα αυτά. Το υπογραμμίσατε ότι η Κομισιόν δεν είναι αυτή που μπορεί να δράσει από μόνη της. Βασιζόμαστε στην προθυμία του Συμβουλίου. Ορισμένες φορές λένε υπογράφουν, αλλά τελικά δεν κάνουν τίποτα άλλο που να υπογράφουν. Ελπίζω πως η Κομισιόν θα τους πιέσει και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα θα ξαναμιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις εισηγήτριες και όσους παρενέβησαν για το ότι ήρθαν εδώ. Λυπούμε για το ότι δεν ήταν τόσοι πολλοί ευρωβουλευτές παρόντες, αλλά υπάρχουν και άλλες ανηλυμένες υποχρεώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι αυτή τη συζήτηση τα κέντρα βάρους και τα θέματα ουσίας που αναφέρατε φυσικά θα τα εντάξουμε στην εργασία μας και θα τα εξετάσουμε με τον ίδιο τρόπο ενδελεχώς και θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα που με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελπίζουμε θα καταλήξουν και θα γίνουν κατανοητά και θα αφομοιωθούν από τους εθνικούς υπαλλήλους των κυβερνήσεων και ε, των κρατών μελών και έτσι συνεισφέρατε σε αυτό. Σας ευχαριστώ όλους και όλες θερμά. Λίγη εδώ η συνεδρίασή μας, η ακρόασή μας. Περνάμε στο σημείο 12. Το έχουμε δει το 13, διάφορα, υπάρχει κάτι υπό τα διάφορα, δεν υπάρχει 14. Επόμενη συνεδρίαση, 15 και 16 Ιουνίου, από τις 3 έως τις 6.30 και από τις 9 έως τις 12.30. Ευχαριστώ όλους τους διερμηνείς, λίγη συνεδρίασή μας, γεια σας.